Bonjour, nous allons commencer notre réunion. Euh, Nous débutons notre réunion par l'adoption de l'ordre du jour. Vous... Καλησπέρα σας. Όπως φαντάζεστε, η επικαιρότητα στην Ουκρανία μας οδηγεί σε αλλαγή της ημερήσιας διάταξής μας, διότι το πρώτο θέμα που προβλεπόταν ήταν κάτι πολύ σημαντικό που είχαμε θέσει από κοινού με την ΕΠΕΞ για την προετοιμασία της διάσκεψης με την Αφρική. Η γραμματεία ήδη το πρωί μας μίλησε για αλλαγή αίθουσας και αλλαγή του πρώτου σημείου. Η ΕΠΕΞ και το καταλαβαίνετε όλοι στις 3 ήθελε λόγω του κατεπήγοντος χαρακτήρα της κατάστασης στην Ουκρανία ιδιαίτερα δε στην Κρυμαία, να αφιερώσει τη συνεδρίασή της στο θέμα αυτό. Προτείνω λοιπόν να αναβάλουμε για τις τέσσερις το σημείο για την προετοιμασία της κοινοβουλικής διάσκεψης κορυφής Αφρικής γιατί το θέμα αυτό δεν θα ζητηθεί πλέον από κοινού με την ΕΠΕΞ αλλά ελπίζουμε ότι ο κύριος Γκάλερο εκπρόσωπός της που προεδρεύει της αντιπροσωπείας με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο θα μπορέσει να έρθει στις 4 γιατί καλό θα ήταν παρουσία του να το συζητήσουμε για να υποφεληθούμε από τις γνώσεις του. Υπάρχει καμία αντίρρηση στην μετατροπή αυτή της ημερήσιας διάταξης. Όχι. Τότε εγκρίνεται με αυτή την τροποποίηση. Λάβατε τα πρακτικά της συνεδρίασης 20-21 Ιανουαρίου. Αν έχετε αντιρρήσεις να τις δηλώσετε στη γραμματεία πριν λήξει η συνεδρίασή μας. Αλλιώς τα πρακτικά θα θεωρηθούν εγκριθέντα. Επίσης λάβατε στους φακέλους σας τις συστάσεις και τις αποφάσεις των συνδονιστών της 11ης Φεβρουαρίου του 2014. Αν έχετε σχόλια για τα συμπεράσματα αυτά, να τα δηλώσετε και αυτά στη γραμματεία πριν λήξει πάλι η σημερινή μας συνεδρίαση, αλλιώς και αυτά τα αποτελέσματα θα εγκριθούν ως έχουν. Έχω μία ανακοίνωση. Γνωρίζετε ότι ήμουν Chief Observer για τις εκλογές στο Νεπάλ και ξαναπήγα μέσα Φεβρουαρίου για την τελική έκθεση με τις συστάσεις μας. Οι συστάσεις αυτές διαπιστώσαμε ότι όλες οι διατάξεις που αφορούσαν την προώθηση της ισότητας των φίλων και των πιο ευπαθών ομάδων δεν είχαν γίνει σεβαστές και άρα ζητήσαμε περισσότερους τέτοιους κανόνες. Επίσης, το εκλογικό σύστημα που αφήνει στα κόμματα τη δυνατότητα να ορίσουν τους υποψηφίους στις ε, αναλογικές εκλογές, συστήνουμε η διάταξη αυτή να καταργηθεί. Υπάρχουν και άλλες τέτοιες ανάλογες συστάσεις, αλλά η αποστολή αυτή κατέληξε πολύ καλά. Το Νεπάλ έχει τώρα κυβέρνηση. Χρειάστηκαν τρεις μήνες για να δημιουργηθεί. Αλλά η εθνοσυνέλευσή τους νομίζουμε ότι θα μπορέσει να εγκρίνει το Σύνταγμα μέσα σε αυτό το έτος. Μήπως η Κομισιόν έχει και αυτή καμία ανακοίνωση να μας κάνει. Όχι, δεν έχει. Δεν λάβαμε κανένα ερώτημα προς την Κομισιόν. Περνάμε λοιπόν τώρα στο σημείο στο σημείο Επτά. Έχουμε την ευχαρίστηση να έχουμε μαζί μας τον κυρίο Ντάμια Έλλη του ΟΣΕΝΤΕΠΕΜ για την παρουσίαση της μελέτης που είχε ζητήσει το Κοινοβούλιο για την εφαρμογή της κοινή στρατηγικής Αφρική-Ευρώπη. Η μελέτη αυτή είναι πολύ επίκαιρη διότι στο τέλος του μήνα στις Βρυξέλλες θα οργανωθεί η διακοινοβουλευτική διάσκεψη Αφρικής Ευρώπης όπου θα συμμετάσχουν πολλοί ευρωβουλευτέ της Επιτροπής μας και έτσι θα μπορέσουμε να αναλύσουμε και καλύτερα ποια μπορεί να είναι η συμβολή του Παναφρικανικού Προγράμματος για τη νέα στρατηγική, ευρωαφρικανική στρατηγική. Ο κύριος Ηλί λοιπόν θα έχει το λόγο για 10 ολόκληρα λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ Θα αρχίσω λίγο στα γαλλικά και μετά θα περάσω στα αγγλικά, μην νομίζετε. Βεβαίω προ μεγάλη μου θλίψη, γιατί είναι και γαλλόφωνη εν μέρη η ε, Αφρικανική Ήπειρο και έχει πολλέ γλώσσε. Αυτό το θέμα τη μετάφραση είναι πολύ σημαντικό στι διεθνεί αφρικανικέ σχέσει. Σα ευχαριστώ πάντω για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μα δίνετε στον οργανισμό μας να παρουσιάσουμε τη μελέτη που μας ε, παραγγείλατε. Donc maintenant, euh, à... Θα περάσω λοιπόν στα αγγλικά γιατί τα έχω στα αγγλικά εδώ. is ε, is a foundation, an independent Είμαστε ένα εξάρτητο ίδρυμα, η CDPM, ερευνητικό κέντρο και εργαζόμεθα ως διαμεσολαβητής στη ε, θέματα διεθνούς συνεργασίας Αφρικής Ευρώπης το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τη Διαχείριση Αναπτυξιακής Πολιτικής, λοιπόν, έχει 50 άτομα προσωπικό περίπου. Εργαζόμαστε σε πολλά θέματα από την επιστημιστική ασφάλεια, διπλωματία, ασφάλεια και ειρήνη, ε, υποδομές ε, και γενικότερα ανάλυση πολιτικής οικονομίας. Εκδίδουμε εκθέσεις ε, και αυτοί που μας παραγγείλατε έχει το τίτλο ε, Rebuilding Confidence and Commitments, επανοικοδόμηση της εμπιστοσύνης και των ε, δεσμεύσεων ε, σε ό,τι αφορά τις σχέσεις Ευρώπης-Αφρικής και την επερχόμενη Σύνοδο Κορυφής. Έχει την εξής δομή λοιπόν η παρουσίαση. Εννέα σημεία. Πρώτον, το πλαίσιο των σχέσεων Ευρώπης-Αφρικής και πώς αυτό μεταβάλλεται δύο θέματα για την εφαρμογή, τα γενικά διδάγματα και ε, επίση τι θα πρέπει να ε, κρατήσουμε από την τελευταία επτά αιτία του ε, Τζάες. Και επίσης ποια είναι η εφαρμογή που λειτουργεί. Το τέταρτο έχει να κάνει με την δομή και την υποδομή με κάποια κριτικά σημεία αναλυτικά. Στη συνέχεια θα έρθω στις παραδοξότητες και τα διλήμματα που έχουμε στη σχέση μας με την Αφρική, ποιες είναι οι προκλήσεις και ποιες δεσμεύσει χρειάζονται από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά χρηματοδότηση της Ένωσης And, uh, και ε, ορισμένες σκέψεις μετά για το πού βρισκόμεθα ένα μήνα πριν την Σύνοδο Κορυφής Ευρώπης Αφρικής της Βρυξέλλες. Και ε, τέλος κάποιες προτεραιότητες για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κάποιες ιδέες για το τι μέλη γενέσθε και πώς ε, θα προχωρήσουν οι σχέσεις μας έτσι, πιο μακροπρόθεσμα. Το πρώτο λοιπόν σημείο. Τι έχει αλλάξει στη σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής. Τι βλέπουμε από πλευράς Αφρικής. Μια νέα αφήγηση, ένα αφήγημα πιο αισιόδοξο ε, με οικονομική άνθηση μια Ήπειρος που αναδύεται και αποκτά περισσότερη εμπιστοσύνη στον εαυτό της, αλλά παραμένουν και πολύ μεγάλες οι προκλήσεις για την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, βιώσιμη ανάπτυξη, ε, σταθερότητα. Υπάρχουν και ζητήματα ε, δημογραφίας τι γίνεται με τις γυναίκες και τους νέους, ποιος ο ρόλος τους. Από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης έχουν αλλάξει τα πράγματα. Πέρασε η κρίση οικονομική, ε, χρηματοπιστωτική αλλά και πολιτική κρίση με όρους Αφρικής και η κρίση στην Ουκρανία επίσης πολύ εύγλωτα σήμερα περιγράφει το γεγονός ότι ε, αστάθεια και απειλές υπάρχουν όχι μόνο στην Αφρική αλλά και στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μάλλον έχει κλονιστεί ως προς την αυτοπεποίθηση και ορισμένοι οι Αφρικανοί μάλιστα τη θεωρούν και μία ήπειρο σε παρακμή. Και το τρίτο είναι η ε, εμφάνιση νέων παγκοσμίων πρωταγωνιστών ε, στην Αφρική που ε, έχουν νέες σχέσεις και συνεργασίες και με τους θεσμούς και με τα κράτη. Έτσι λοιπόν έχει το πλαίσιο για το επόμενο διάστημα και για την επόμενη σύνοδο κορυφής. Ποια είναι λοιπόν τα διδάγματα που μπορούμε να εξακάκουμε από την εφαρμογή του Τζάις που είναι και ε, πολιτική ε, εξαγγελία, θέλετε και πρόγραμμα. Τι μπορούμε λοιπόν να συναγάγουμε. Θα πρέπει να καταλάβουμε το εξή. Οι οχτώ εταιρικέ σχέσεις ε, έχουν αναπτυχθεί αυτόνομα με το δικό τους ρυθμό και το δικό τους τρόπο με μεγάλη ποικιλία διαλόγων και τρόπων εφαρμογής. Ε, οι θεματικές εταιρικές σχέσεις και ενότητες είχαν συμπροέδρους. Και όποτε αυτοί επέλεγαν φάνταστες και ευέλικτες ε, εφαρμογές, ε, είχε αποτέλεσμα αυτό και απέδιδε. Και το πλαίσιο αυτό ήταν πάρα πολύ υποστηρικτικό για το διάλογο. Το αντίθετο όταν συνέβαινε, απροθυμία ακινησία εμπλόκαρε τη συνεργασία και το διάλογο. Και αυτό ισχύει πάρα πολύ ε, συμφωνίες ε, οικονομικής συνεργασίας στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ή ε, μίζωνες ε, κρίσεις ασφαλείας. Λοιπόν, ας δούμε λίγο πιο κοντά την προηγούμενη εφαρμογή, την ευέλικτη και φάνταστη. Σε ό,τι αφορά τις υποδομές ασφάλειας και ειρήνης, Ε, ο διάλογος ε, υποστηρίχθηκε πάρα πολύ από χρηματοδότηση που υπήρχε στο παρελθόν και επεκτάθηκε πέρα από το ε, περιορισμένο πλαίσιο του τζάις στην περιφερειακή ολοκληρωσή και στο εμπόριο είδαμε ότι από τη μια είχαμε τις διαπραγματεύσεις για τις εμπορικές συμφωνίες και από την άλλη ε, το κέντρο αυτό, το Τζάες, και είπαν ορισμένοι ενεχόμενοι στο δεύτερο εγχείρημα ότι η συμφωνία ΣΕΠΑ ήταν ένα καλά σχεδιασμένο ε, πολιτικό και οικονομικό καταστροφικό πρόγραμμα. Επίσης, οι επιμέρους Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ασχολήθηκαν με θέματα επιμέρους ε, ο διάλογος στα ανθρώπινα δικαιώματα και ε, στη δημοκρατική διακυβέρνηση ήταν σκληρός κατά τη διάρκεια των ετών. Βρέθηκαν κάποιες εφάνταστες και πάλι λύσεις και στην πολιτιστική συνεργασία ε, ως προς ε, τη Σύνοδο Κορυφής εδώ αναφέρομαι στην Καζαμπλάνκα για το λαθρεμπόριο πολιτιστικών αγαθών. Επίσης, ε, σε θέματα επιστήμης, κοινωνίας των πληροφοριών και διαστήματος ε, έχει ενταθεί η συνεργασία, ιδιαίτερα προς το διάστημα. Αν θέλετε θα πω και σε λεπτομέρειες Τώρα, τι κάνει κανείς με τη διαρθρωτική, μάλλον τη θεσμική διάρθρωση. Είναι βαριά, αλλά έχει μόνο συμβουλευτικό χαρακτήρα. Και προσπαθήσαμε να ε, κάνουμε ένα διάγραμμα, μια γραφική παράσταση που ε, θα σας έδειχνε πόσο περίπλοκη είναι αυτή η δομή. Ακόμα και αν δεν βλέπετε τις λεπτομέρειες, είναι εύγλωτη η εικόνα που αντικρίζεται στην οθόνη. Ε, καταλήξαμε ότι δεν μπορεί να υπάρχει ένα μοντέλο για όλες τις καταστάσεις, δεν προσφέρεται αυτό. Η εφαρμογή ακόμα δεν έχει αξιολογηθεί σωστά. Δεν υπάρχει αρχή της επικουρικότητας και δεν ξέρουμε σε ποιο επίπεδο θα πρέπει να είναι η συνεργασία. Σε ε, υπηρετικό, περιφερειακό, εθνικό, τοπικό, όλα αυτά μαζί. Και ε, το επόμενο συμπέρασμα ε, της μελέτης είναι ότι η δομή αυτή δεν συνδεόταν με τα πραγματικά κέντρα λήψεων αποφάσεων ούτε στην Αφρική ούτε στην Ευρώπη. Τώρα τι γίνεται, παραμένουν κάποια παράδοξα και κάποια διλήμματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και να λυθούν είτε κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής είτε αργότερα, εάν θέλουμε να είναι καλής ποιότητας η συνεργασία και να παραμείνει. Το πρώτο, υπάρχει πρόβλημα, έλλειμμα ηγεσία εκατέρωθεν. Identify... Ε, ήταν πολύ δύσκολο να καταλάβουμε ποιοι είναι οι εκπρόσωποι, οι διαπραγματευτές. Ε, ε, ήταν συγκεχημένη η εικόνα. Δεν υπήρξε καμία υπουργική ε, συνέντηση από το 2010 και μετά. Δηλαδή έχει χάσει την πολιτική ορμή αυτό το και, και η καθοδήγηση το εγχείρημα. Μετά έχουμε βαριά υποδομή εφαρμογής όπως είδαμε προηγουμένως, πράγμα που δημιουργεί εντάσεις. Από τη μια καταβάλλονται προσπάθειες για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και από την άλλη είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε τη δεδομένη αρχιτεκτονική. Ένα τρίτο παράδοξο είναι η ασυμμετρία. Όταν ακούμε το αφήγημα για ε, ε, επίσης όρης ε, σχέση, βλέπουμε συμμετρίες και στις ικανότητες και στις δυνατότητες μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής. Λοιπόν, μεγάλες εντάσεις και μεγάλες ασυμμετρίες. Επίσης, μονομερής ο σχεδιασμός από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη μια και της χρηματοδότησης και από την άλλη το πνεύμα της συνεργασίας και στην χρηματοδότηση. Επίσης έχουμε και συγκρούσεις στην ε, χρηματοδότηση. Υπάρχουν χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά δεν υπάρχουν από την Αφρική για τη συνυπευθυνότητα ή συγχρηματοδότηση. Αυτά είναι τα συμπεράσματα μετά από μία επταετία εφαρμογής. Ας έρθουμε τώρα στην κοινωτική χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε. της ε, κοινή στρατηγικής οι ε, χρηματοδοτικοί μηχανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάρα πολύ περίπλοκοι. θα πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι δημιουργήθηκε το Παναφρικανικό Πρόγραμμα ε, μέσα στο DCI. Και θα πρέπει να το δούμε αυτό στην επόμενη φάση εφαρμογής του μέσου αναπτυξιακή συνεργασίας. Καθώς βαίνουμε λοιπόν προς τη Σύνοδο Κορυφής, το βασικό μήνυμα της μελέτης είναι ότι ακόμα υπολοιπόμεθα ως προς τη φιλόδοξο πολιτικό όραμα και τη διακήρυξή του. Θα πρέπει και οι δύο πλευρές να διατρανώσουν και πάλι την προθυμία τους για την κοινή συνεργασία την οποία εμπνεύστηκαν το 2007. Θα πρέπει να αναζωογονηθεί και ανοικοδομηθεί και η εμπιστοσύνη και οι δεσμεύσεις. Έχουν γίνει κάποιες κινήσεις για να ξεπεραστούν τα εμπόδια, ανθρώπινα δικαιώματα, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, προσκλήσεις Αφρικανών ηγετών, όλα αυτά συστηματικά ε, τα ε, εξέταζαν ε, και εν ώψη της Συνόδου Κορυφής κάθε φορά και θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Αλλά υπάρχουν τώρα δύο τινά. Μία κάπως πιο light σύνοδος κορυφής με λιγότερες φιλοδοξίες ή περισσότερες προσπάθειες για να υπάρξει πολιτική ηγεσία και στα κοινοβούλια και να είναι αυτή η συνεργασία και η στρατηγική πιο ενδιαφέρουσα σε πολιτικό επίπεδο. Τι έχουμε λοιπόν να προτείνουμε στο Κοινοβούλιο τώρα ως συστάσεις. Έχουμε εντοπίσει τρεις ε, τομείς που χρειάζονται περισσότερη προσοχή. Το πρώτο είναι το πολιτικό επίπεδο και πολιτικές διακήρυξεις. Θα πρέπει να είναι πιο διάκριτη η ε, πολιτική καθοδήγηση. Ποιος κάνει κουμάντο, ας πούμε, ποιος έχει το γενικό πρόσταγμα. Πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις ε, για τη χρηματοδότηση και ποια είναι η μακροπρόθεσμη στρατηγική για την Ευρώπη και την Αμερική. Θα πρέπει επίσης να ε, δούμε και σε ποιο επίπεδο επεμβαίνει η επικουρικότητα στην Αφρική. Το δεύτερο, ποιότητα διαλόγου και εφαρμογή. Γίνονται προσπάθειες για να συνδεθούν ε, οι δομέ λήψη αποφάσεων και στην Ευρώπη και στην Αφρική και προσπαθείς να δημιουργηθεί περισσότερος χώρος για διάλογο ε, έτσι, σε επίπεδο άτυπο συμπεριλαμβανομένης και της κοινωνίας των πολιτών και των διαφόρων ενδιαφερομένων. Και το τρίτο στοιχείο είναι ο έλεγχος, η εποπτεία, η ενίσχυση των μηχανισμών και να οριστείτε καλύτερα ο ρόλος των κοινοβουλίων σε όλο αυτό το εγχείρημα. Τώρα, κάποιοι προβληματισμοί για σας, για την Επιτροπή σας και τη συνεδρίασή σας για το μέλλον. Ίσως πρέπει να δούμε και το θέμα των οτροπιών, των στάσεων, των συμπεριφορών, των αντιλήψεων. Ποιο είναι το αμοιβαίο συμφέρον μας η Αφρική επίσης είναι ε, ένας τόπος ευκαιριών και θα πρέπει να το καταλάβουμε. Πώς μεταφράζεται αυτή η νέα πραγματικότητα σε διπλωματική συνεργασία και ευρύτερες ε, Ποιες είναι οι εμβληματικές ε, πρωτοβουλίες που θέλουμε να ξεχωρίσουμε. Οι Ευρωπαίοι έχουν καταλάβει ποια είναι τα στρατηγικά του συμφέροντα στην Αφρική. Και επίσης η Αφρική είναι ένα ενιαίο σύνολο. Και ποιος θέλει να θεωρείται ένα μπλοκ η Αφρική, ένα μπλοκ η Ευρώπη. Και μετά, τι μέλη γενέστε, αυτό είναι πιο μακροπρόθεσμο, μετά τη λήξη της συμφωνίας του Κοτονού το 2020. Και αυτό χρειάζεται σκέψη και ίσως από κοινού θεώρηση όπου η κάθε πλευρά θα κάνει τα μαθήματά της, για να το πω έτσι, ε, για το νέο τρόπο συνεργασία. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν επιθυμεί να κάνει ερωτήσεις. Και στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, ο κύριος Ζωσέ Κώστα Περέρα. Um, Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Μπορούμε να συμφωνήσουμε στα όσα ο καλός φίλος μόλις σας παρουσίασε σήμερα. Αναφέρθηκε στα κυριότερα θέματα που καλύπτουν την κοινή εταιρική σχέση και για τη στρατηγική μεταξύ Ευρώπης Αφρικής και τα ανέφερε και σε σχέση με τις μεγάλες φιλοδοξίες πολιτικής ε, στρατηγικής αυτή την εταιρική σχέση μεταξύ των φορέων και υπηρεσιών πρέπει να επαναθεωρηθούν και να βελτιωθούν όλα αυτά για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Το μόνο σημείο που δεν θα ήμουν τόσο βέβαιος όπως είναι εκείνο είναι εκεί όπου ταυτοποίησε, εντόπισε στις ε, μικτές ε, ομάδες πραγματονομών ε, την επαρκή δημιουργικότητα λέει από πλευράς προτάσεων σαν συνέπεια της ε, σύμπτωσης ε, των ε, μελημάτων των δύο πλευρών για το όσο, όσα πρέπει να γίνουν πρέπει να μπορούν να στεφθούν με κάποιο βαθμό επιτυχίας πρέπει να στραφούμε και να δούμε με διαφορετικό τρόπο τη μορφή αυτή κάποιο τρόπο που θα λαμβάνει υπόψη όχι μόνο το επίπεδο φιλοδοξίας αλλά και άλλους παράγοντες όπως το δυναμικό, την δυνατότητα να ανταποκριθούμε στις προϋποθέσεις και τις χρηματοοικονομικές συνθήκες και όρους πρέπει να συγκλίνουμε σε σχέση με την ίδια την πραγματικότητα στις δράσεις μας αυτές. Αυτό είναι εκείνο το οποίο σχεδιάζουμε να κάνουμε και αυτό σχεδιάζουμε να κάνουμε κατά τη διάρκεια της επόμενης συνόδου κορυφής, να εμβαθύνουμε σε αυτά τα θέματα με τους Αφρικανούς εταίρους ώστε μια και εκείνοι έχουν και εκείνοι επικρίσεις και κριτικές παρατηρήσεις σε αυτό το κοινό πρότυπο. Για το ότι συμφωνούμε για τη διάγνωση δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε και για τη θεραπεία. Υπάρχει λοιπόν διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά την οπτική γωνία. Το να συμφωνήσουμε λοιπόν ότι τα πράγματα όπως είχαν δεν μπορούν να συνεχιστούν είναι ήδη κάτι πολύ θετικό. Ανέφερε κάποια σημαντικά θέματα όπως ε, ιδιαίτερα το σημείο εκείνο για τις προκλήσεις και τα διλήμματα τα οποία αντιμετωπίζουμε, παράδοξες κατα... Ε, καταστάσεις που κάποια από αυτά τα προβλήματα δεν θα μπορέσουν να επιληθούν ούτε στη Σύνοδο Κορυφής ούτε στους επόμενου μήνε και χρόνια. Παίρνει πολύ χρόνο. Μία ολόκληρη γενεά, για παράδειγμα, χρειάζεται χρονικά για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε αυτές τις δράσεις στο βαθμό εκείνο όπως αναμένουμε να μπορέσει να επιτευχθεί αποτελεσματική δράση. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν, είναι, δεν ε, παραλληλίζονται και αντιστοιχούν υποχρεωτικά με την ίδια την πραγματικότητα. Είναι το θέμα λοιπόν του προτύπου εφαρμογής, αναθεώρησής του. Καλή ευκαιρία να ξαναπροβληματιστούμε γι' αυτό και να δούμε αυτό το οποίο επισημάθηκε, δηλαδή για τους δικούς μας στρατηγικούς στόχους και τους αφρικανικούς στρατηγικούς στόχους. Να μπορέσουμε να βρούμε έναν τρόπο συγχρονισμού μεταξύ τους, ώστε να είναι θετικά τα αποτελέσματα του συσχετισμού μεταξύ των δύο υπήρων της Ευρώπης και της Αφρικής. Επίσης θα ήθελα να υπογραμμίσω μια παρατήρηση που έκανε για την ανάγκη η κοινωνία των πολιτών να εμπλακεί, να είναι μέρος αναπόσπαστο αυτής της στρατηγικής. Η στρατηγική πρέπει να έχει στο επίκεντρο τους ανθρώπους όμως η πραγματικότητα είναι ότι οι οργανώσεις και οι οργανισμοί της κοινωνίας των πολιτών δεν έχουν επιτύχει το επίπεδο το ευκταίο το οποίο θα επιθυμούσαμε να υλοποιηθεί. Πρέπει να δούμε λοιπόν ποιος θα είναι ο ρόλος του σε οποιαδήποτε διατύπωση συμφωνηθεί μεταξύ των δύο πλευρών. Θα πρέπει να επαγρυπνούμε λοιπόν ώστε η κοινωνία των πολιτών να έχει πραγματικά ένα ρόλο να διαδραματίσει. Τώρα, μηχανισμοί εποπτείας, μηχανισμοί διαφάνειας, μηχανισμοί παρακολούθησης, follow-up για το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα αυτού του κοινού έργου όσον αφορά ε, πραγματογνώμονες σε τεχνικό επίπεδο είναι κάτι το οποίο καλωσορίζουμε και είναι και αναγκαίο πρέπει να μπορέσουμε να το πετύχουμε χωρίς να δημιουργήσουμε μια άλλη, ένα άλλο διάστρωμα γραφειοκρατικού βάρους και γραφειοκρατικής επιβάρυνσης που θα αυτοτροφοδοτείται μεν αλλά δεν θα επιτυγχάνει τον στόχο που θέλουμε να επιτευχθεί. Πρέπει λοιπόν αυτή η ανάγκη να ληφθεί υπόψη, να επαγρυπνούμε και να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Σίγουρα και για το ρόλο του Ευρωκοινοβουλίου επίσης που πρέπει και αυτό να συμμετέχει στην διαδικασία εποπτείας και επιτήρησης και ελπίζω ότι θα υπάρχει το δυναμικό να αυξηθεί ο διάλογος αυτός, η συνιστόσα του διαλόγου με το Ευρωκοινοβούλιο για τη συνεργασία μας για να μπορέσουμε αυτούς τους κοινούς στόχους να τους επιτύχουμε από κοινού. Συνολικά σφαιρικά λοιπόν νομίζω είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ καλή προσπάθεια αυτό το εγχείρημα στρεφόμενοι προς το μέλλον. Και όχι μόνο αυτό, αλλά επίσης Θέλω να δώσω και επένους στον Ντάμιεν για το καλό έργο που έχει επιτελεστεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Μαρτίνες τώρα. Ευχαριστώ συνάδελφε πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω για την παρουσίαση που μας έγινε και πιστεύω ότι είναι ενδιαφέρουσα και επιπλέον είναι επακριβέστατη μέσα στους περιορισμούς που θέτει ο χρόνος και η εμπειρία που έχουμε ακριβώς εμείς δεν είναι ακριβώς εκείνη για το ότι πολλές από τις προσωπικότητες και φίλους που έρχονται να παρουσιάσουν ένα έγγραφο τέτοιας φύσης είναι ικανοί πραγματικά να συνοψίσουν τα πράγματα τόσο αποτελεσματικά όπως το έκανε αυτός που μας παρουσίασε αυτά τα θέματα σήμερα εδώ. Έχω δύο-τρία σχόλια να κάνω, όχι τόσο σε σχέση με αυτά που μας αναφέρθηκαν, αλλά για την γενικότερη προβληματική, με δύο-τρεις διαφοροποιήσεις που πρέπει να τις δούμε γιατί θα έχουν επιπτώσεις φυσικά στην κοινοβουλευτική σύνοδο που θα έχουμε κατά τα τέλη του μήνα. Πρώτα απ' όλα λοιπόν πιστεύω ότι υπάρχει μια ερώτηση που τίθεται για το αν η Αφρική είναι μία ή δεν είναι μία και ενιαία. Και φυσικά στη συνέχεια για την προσέγγιση και τοποθέτηση που υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωκοινοβούλιο σε σχέση με την Αφρική μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Κάνουμε λόγο για δύο Αφρικές. Την Μεσογειακή Αφρική αφενός και αφετέρου για την υπόλοιπη, λυπή Αφρική. Αυτό τίθεται κάθε φορά με όλο και περισσότερο οξυμένο πρόβλημα σε σχέση με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο ε, υπάρχει ένα πρόσθετο στοιχείο όπως το γεγονός αυτό και που πάλι βλέπουμε το ίδιο πρόβλημα να υφίσταται σε σχέση με τις σχέσεις με την Αφρικανική Ένωση. Και αυτό γιατί. Γιατί πρώτον, μέσα από όλο αυτό το έργο και προοπτική συνεργασίας υπάρχει αυτός ο κατακαιρματισμός σε δύο διαφορετικές υπήρους, με δύο διαφορετικούς εταίρους, με δύο διαφορετικές προβληματικές και όταν συναντώμεθα με την Αφρικανική Ένωση ή το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο δεν συναντώμεθα με δύο αλλά με ένα. Αλλά αυτό είναι ένα πρόβλημα, ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το προαγάγουμε και να προχωρήσουμε πέρα από το πρόσθετο στοιχείο που απορρέει από το ότι η Αφρικανική Ένωση και η Αφρική δεν είναι μόνο το Μαρόκο για παράδειγμα ε, εταίρος που είναι ξεχωριστός εταίρος σίγουρα αλλά αναντικατάστατος κιόλας και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την άλλη πλευρά γνωρίζουμε ότι για συγκεκριμένους λόγους που όλοι γνωρίζουμε, ιστορικούς λόγους κτλ, βρισκόμαστε στο ότι στην Αφρικανική Ένωση υπάρχει άλλος εταίρος, υπάρχουν άλλοι εταίροι απέναντί μας, που παρότι υπάρχει αυτό το πλαίσιο, το ξεχωριστό πλαίσιο το οποίο αντιμετωπίζουμε με ιδιαίτερη προσοχή, παρόλα αυτά δημιουργείται μια δυσλειτουργία. Ήδη το ίδιο το όνομα, ο τίτλος των σχέσεών μας δεν είναι οι σχέσεις ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρικανική Ένωση, αλλά η σύνοδος είναι η σύνοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική. Τελεία και παύλα. Και αυτό είναι ένα πρώτο πρόβλημα που δεν μπορούμε και να το αγνοήσουμε καθόλου. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει και ένα θέμα πιο συγκεκριμένο, πιο εξειδικευμένο, που φοβούμε ότι θα μπορούσε να μας να αναλώσει όλη την προσπάθεια στην Σύνοδο Κορυφής. Ένα πρώτο πρόβλημα είναι το θέμα το ότι δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι κατά τα τελευταία τρία ή τέσσερα χρόνια ζήσαμε, βιώσαμε ένοπλες σειράξεις, σοβαρότατες και βαρύτατες σε διαφορετικές αφρικανικές χώρες. Φυσικά όλοι συγκινούμεθα για την κατάσταση στο Μάλι για παράδειγμα, για την κεντροαφρικανική δημοκρατία επίσης. Αν δούμε όμως λίγο πιο πίσω το τι συνέβη σε μια ανασκόπηση, αυτό που έγινε στην ε, ε, Μεσογειακή Αφρική πάλι είχαμε πράγματα τα οποία συνεπαγόντουσαν, για παράδειγμα το τι συνέβη στην Λιβύη και συνειδητοποιούμε ότι αυτές οι σειράξεις είναι σειράξεις που δεν κλείνουν δεν επουλώνονται αυτές οι ουλές αλλά συνεχίζουν να είναι ανοιχτές και να πιωροούν και να υπάρχουν προβλήματα εκεί και ζούμε μια ας το πω έτσι οδυνηρή έκπληξη στη Λιβύη για παράδειγμα τις τελευταίες 48 ώρες κιόλας για να μην πάμε και πιο μακριά το τι γίνεται εκεί Λοιπόν, βλέπουμε ποια είναι η πραγματική κατάσταση που δημιουργείται και ποια κατάσταση έχουμε μπροστά μας εκεί. Και για το Μαλί ας ελπίσουμε ότι θα είμαστε πιο ικανοί να συνεισφέρουμε να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα. Το τελευταίο πρόβλημα που θέλω να αναφέρω, που θα είναι αναπόφευκτο, διότι αφορά και την ε, Ευρωβουλή μας και μέλη της ομάδας μας που θα θέσουν προτεραιότητα σε αυτό το θέμα είναι η κατάσταση η οποία είναι πραγματικά σύμβατη και απαράδεκτη με τη μορφή σχέσεων που μπορεί να αναπτύσσει και να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτές τις χώρες, για παράδειγμα την κατάσταση στην Ουγγάντα, όχι μόνο την ομοθεσία και κατάσταση στην Ουγγάντα, την καταδίωξη δηλαδή τους διωγμούς, διωγμούς όσον αφορά το φύλλο, δηλαδή όσον αφορά τους ομοφιλόφιλους, την ιδιότητα του ομοφυλόφιλου σε αυτή τη χώρα διωγμή και καταπίεση. Επί μια ολόκληρη σειρά ετών προσπαθήσαμε να το αντιμετωπίσουμε. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα το οποίο το θυμάμαι στις συνόδους κορυφή, ε, των χωρών ΑΚΕ. Προσπαθήσαμε να προχωρήσουμε σε αυτό το πεδίο. Είναι όμως προφανές ότι η κατάσταση οπισθοδρόμησε, ε, σημείωσε μια πραγματικά δραματική οπισθοδρόμηση και το βλέπουμε αυτό και σε σχέση και με τα κείμενα. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν σε αυτή τη συνάντηση που θα έχουμε αυτό το θέμα να μην είναι ένα θέμα το οποίο θα τεθεί στο Προεδρείο και, θα, και δεν μπορεί να μην μας απασχολήσει. Διαφορετικές κοινοβουλευτικές ομάδες βλέπουμε ότι δεν μπορούν να προσεγγίσουν τις σχέσεις με τις αφρικανικές χώρες χωρίς να θέσουν πραγματική προτεραιότητα σε αυτό το πρόβλημα, σε αυτό το θέμα. Τώρα δεν ξέρω πώς οι πραγματογνώμονες και οι ε, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βλέπουν και αντιμετωπίζουν την κατάσταση που θα έχουμε μπροστά μας και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Δεν θα υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα σε μια τόσο ξεχωριστή στιγμή σε αυτή τη σύνοδο κορυφής. Ε, λοιπόν τι θα δούμε. Θα δούμε ότι για μια χώρα σαν την Ουγγάντα και γύρω από αυτό μπορεί να υπάρξει το ότι αν δεν είμαστε ευφυείς και φάνταστοι στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, μπορεί να υπάρχει μια ένωση Αφρικανών, Αφρικαν, ε, Αφρικανικών χωρών που δεν είναι τόσο κοντά στις, στις θέσεις της Ουγγάντα από πλευράς νομοθεσίας της Ουγγάντα και όχι μόνο στην νομοθεσία τους αλλά και τις δηλώσεις και τοποθετήσεις δημόσιες του Προέδρου που είναι προκλητικές κιόλα θα έλεγα βρίσκονται στο όριο της προκλητικότητας λοιπόν θα ήθελα από πλευράς της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης και από πλευράς των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μας πούν, να μας έλεγαν πώς βλέπουν και πώς διαμορφώνεται αυτή η προβληματική σε σχέση με τις σχέσεις μας με τις αφρικανικές χώρες, την Αφρική και τις ε, χώρες στις οποίες αναφέρομαι. Διότι δεν πιστεύω ότι μπορεί να έχουμε κάποιο συμφέρον, να έχουμε μια σύνοδο κορυφής η οποία θα ε, τερματιστεί, ας το πω έτσι, μέσα σε κενό χωρίς να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να ανοίξουμε τα θέματα ουσίας. Και γι' αυτό λοιπόν αυτό το θέμα δεν θα μπορέσουμε να το αποφύγουμε, δεν θα μπορέσει να αμεληθεί και σαν συνέπεια των τοποθετήσεων ε, κάποιων από τις ομάδες μας και είναι και δικαιολογημένο αυτό. Είναι απόλυτα δικαιολογημένη αυτή η τοποθέτηση. Ευχαριστώ πρώτα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε αυτή τη στιγμή θέλω και εγώ να δραχθώ της ευκαιρίας οπωσδήποτε για να το αναφέρω αυτό. Η έκθεση αυτή είναι πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση. Θέλω να ευχαριστήσω για την έκθεση αυτή και για το πώς θα μπορούσε κανείς να πει και να διαμορφώσει το ότι οι σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, ε, Αφρικής ε, έχουν πάρει αυτή την τροπή με τον διπλωματικό έστω αυτό τρόπο είναι σίγουρο ότι απευθύνεται έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωκοινοβούλιο και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ώστε να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη και να αποκαταστήσουμε τις δεσμεύσεις μας και από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης το είπε και θα πρέπει να ενδυναμωθούν αυτές οι σχέσεις ε, του ρόλου μας ε, στην Αφρική και πρέπει να επανεξετάσουμε και να επαναξιολογήσουμε τι κάνουμε στην Αφρική και πώς θα θέλουμε να προχωρήσουμε. Είναι ένα θέμα το οποίο σχολίασε και ο συνάδελφος Μιγελάνχελ Μαρτίνεθ. Λοιπόν, το Ευρωκοινοβούλιο κάνει συνεδριάσεις και αυτή και όλα στη χρονική στιγμή με τις διάφορες ε, ομάδες του για να υπάρξει η διαμόρφωση αυτού του στρατηγικού διαλόγου για αυτά τα θέματα και σε σχέση με την Παναφρικανική ομάδα και θα γίνει λόγος ε, για αυτά τα θέματα και πρέπει το Ευρωκοινοβούλιο να τοποθετηθεί για αυτά τα θέματα και συγκεκριμένα για αυτό το θέμα που αναφέρθηκε πιο πριν. Θέλω να δραχθώ αυτή τη ευκαιρία για να γνωρίζω ποια είναι η άποψή σας, να μάθω ποια είναι η άποψή σας για την ανάπτυξη, για τους στόχους της χιλιετίας, ε, την, τους στόχους της χιλιετίας, ένα θέμα το οποίο πρέπει παράλληλα να επικεντρωθούμε σε αυτό σε σχέση με την ανάπτυξη των σχέσεων μας με τις χώρες της Αφρικής. Είναι πολύ σημαντικό και για την χώρο την βιώσιμη ανάπτυξη, το θέμα της ασφάλειας. Και γι' αυτό που ε, έκανε λόγο ο συνάδελφος Μιγελάνχελ Μαρτίνεθ είναι θεμελιώδους σημασίας να δούμε πώς από την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να έχουμε μια σαφή και καθορισμένη δεδομένη στρατηγική για τα θέματα της ασφάλειας στην Αφρική και στην Ουκρανία ζήσαμε πρόσφατα στο μια κατάσταση όπου κανείς δεν είχε προβληματιστεί το τι θα μπορούσε να γινόταν λίγο πιο πέρα στο μέλλον. Λοιπόν, να δούμε το θέμα αυτό σε μια τέτοια προοπτική, να αναπτυχθεί μια σαφής ε, ε, δεδομένη στρατηγική από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από το Ευρωκοινοβούλιο, φυσικά για να υπάρξει εμπιστοσύνη και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε σχέση με τα όσα ανέφερε ο ε, φίλος και εταίρος μας και να ακούσουμε ποια είναι η άποψή σας για αυτό το θέμα. Και μια ερώτηση. Όλοι ξέρουμε ότι βλέπουμε μια αλλαγή και στον τομέα της συνεργασίας με νέους εταίρους και με το ιδιωτικό κεφάλαιο όσον αφορά τη συνεργασία. Και αυτό πάλι μπορεί να αποτελεί μια ευκαιρία. Θα ήθελα και πάλι να μας πείτε την άποψή σας. Ποια είναι η θέση σας, ποια είναι η θέση της Επιτροπής ε, σε σχέση με αυτές τις σχέσεις, με αυτή τη σχέση. Γιατί και το ιδιωτικό κεφάλαιο μπορεί να είναι μια ευκαιρία την οποία πρέπει να, χρησιμο... να εκμεταλλευτούμε για τη μέγιστη διαφάνεια, να δούμε θα... Ε, ποιες επιπτώσεις θα υπάρξουν μέσω ε, αυτών των δράσεων στις διμερείς σχέσει. Συμφωνώ είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση που ε, εφιστά την προσοχή στα θέματα αυτά σε σχέση με το συσχετισμό της Ευρώπης με την Αφρική για αυτή τη στρατηγική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ελή, σας ξαναδίνω το λόγο για να απαντήσετε στις ερωτήσεις των βουλευτών, στις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. και τους κυρίους βουλευτάς για όσα είπαν και σχολίασαν. Θα πάρω τις ερωτήσεις μία-μία, αλλά είναι πολλές. Για τη γενική διάγνωση, δηλαδή, πώς να χαρακτηρίσουμε τις σχέσεις των δύο υπήρων. Πριν από ένα χρόνο είχα γράψει σε ένα άρθρο για το περιοδικό του Ιδρύματος της Νότιας Αφρικής ε, Διεθνών Σχέσεων με τίτλο ίσως λίγο απεσιόδοξο σήμερα έλεγε τα σφάλματα στην απομάκρυνση των υπήρων. Υπήρχε δηλαδή κίνδυνος απομάκρυνσης των δύο υπήρων μεταξύ τους, αλλά και κατακρίμνησης της κάθε μίας ρήγματος. Οι προσπάθειες που γίνονται σήμερα για την προετοιμαστή διάσκεψη δείχνουν ότι υπάρχουν παράγοντες που θέλουν να αποφύγουν την απομάκρυνση, αλλά για να αποφευθεί και το ρήγμα δεν έχει γίνει τίποτα. Το θέμα λοιπόν είναι ποιες είναι οι σχέσεις ε, μεταξύ εκείνων που θέλουν σύγκληση και εκείνων που δεν ενδιαφέρονται για αυτήν. Μια πιο λεπτομεριακή ανάλυση της θέσης των διαφόρων παραγόντων χρειάζεται και γι' αυτό έρχομαι στο ερώτημα για τη διαφορά <laughs> μεταξύ Νότιας Αφρικής και υπολείπου Αφρικής. Ξέρουμε ότι υπάρχει αυτό το spaghetti bowl των περιφερειακών αφρικανικών οργανώσεων ότι υπάρχουν περιφερειακές δυνάμεις στην Αφρική που δεν χρειάζονται μάλλον τις περιφερειακές αυτές οργανώσεις αλλά τις χρησιμοποιούν μόνο όταν τους βολεύει. Κάτι ανάλογο ισχύει και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη-μέλη που είναι αρκετά ισχυρά και μπορούν να δράσουν μόνο τους το πράττουν. Όταν χρειάζονται και τους άλλους επανέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να εξευρωπαίσουν σε εισαγωγικά ορισμένα στοιχεία της πολιτικής τους. Είναι λοιπόν μια διαλεκτική πολύ κινητική και το θέμα είναι πώς να εκμεταλλευτούμε όλες τις ευκαιρίες για συνεννόηση και εμπιστοσύνη αν υπάρξει μια πρωτοβουλία κάποιου αφρικανικού ή ευρωπαϊκού κράτους που καταλήγει σε μεγαλύτερη σύγκληση των δύο υπήρων, γιατί όχι. Αλλά πάντως για το jazz νομίζω ότι το θέμα της επικουρικότητας είναι πολύ σημαντικό. Και η πυρωτική διάσταση, η δημιουργία του Πανάφ, είναι κάτι ιστορικής σημασίας, καινούριο, και μάλλον αυτό θα δημιουργήσει τελικά τη διαφορά αν οι συζητήσεις για τη χρήση των ταμείων του γίνουν με εμπιστοσύνη γιατί ένα από τα βασικά σημεία της εταιρικής αυτής σχέσης είναι η χρηματοδότηση. Αυτή τη φορά θα υπάρξει. Δεν θα υπάρχει πια δηλαδή η δικαιολογία ότι δεν έχουμε λεφτά αλλά πρέπει να υπάρξει συνεργασία για... με αυτό το πνεύμα. Είναι μια προσπάθεια που πρέπει να γίνεται συνεχώς. Η προσωπική μου θέση πάντως είναι ότι η πυρωτική διάσταση πρέπει να τονιστεί όταν μιλάμε για το GED Και τα υπόλοιπα επίπεδα, εθνικό, περιφερειακό, όπου υπάρχουν δεκάδες χιλιάδων προγράμματα, δεν χρειάζεται να συζητηθούν από το τζιάδ. Αυτό όμως προσωπικά. Τώρα για τις διανέξεις και διαμάχες. Δεν επέμεινα μεν, αλλά η ποιότητα της συνεργασίας και στο θέμα της ειρήνης και της ασφάλειας είναι εξαιρετική μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής. Πήγα στην Αντίσα Μπέμπα τον Νοέμβριο για να συνεννοηθώ με εκπροσώπους της Ένωσης που είναι υπεύθυνοι για την ειρήνη και την ασφάλεια και τους αντίστοιχους αξιωματούχους της Αφρικανικής Ένωσης και όλοι έχουν συνέστηση της ποιότητας της συνεργασίας αυτής. Υπάρχει ένα κοινό άραμα, εμπιστοσύνη, πόροι και συγκεκριμένα επιτεύγματα. Δέστε τη Σομαλία. Δέστε τι γίνεται σήμερα στο Σαχέλ. Η Αφρικανική Ένωση παίζει όλο και σημαντικότερο ρόλο και ο διάλογος με την Ευρώπη είναι πολύ καλός. Είδεστε τι ποιότητα ήταν η διάσκεψη του μεγάλου των Ηλυσίων για την Αφρική. Νομίζω ότι εδώ έχουμε ένα παράδειγμα επιτυχίας και κοινού οράματος. Υπάρχουν πολλοί βέβαια τρόποι να πραγματοποιηθεί αυτό. Ο Γαλλικός όταν η Γαλλία παρεμβαίνει μόνη της ή και με άλλους, ο Αφρικανικός τρόπος όπως στη Σομαλία και υπάρχουν και ευρωπαϊκοί τρόποι όπως με το φορκά. Το αφρικανικό τρόπος χρειάζεται περισσότερο χρόνο για εφαρμοστή αλλά προοδεύει. Που είμαστε σε μεταβατική περίοδο που αλλάζουμε τρόπους. Όσο δεν υπάρχουν μεγαλύτερες δυνατότητες για την Αφρική θα χρειάζεται περισσότερη ευρωπαϊκή βοήθεια αλλά θα δούμε αν τελικά η απάντηση που πρέπει να δοθεί είναι συλλογική, εθνική ή όχι. Πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα ευέλικτα λοιπόν, αλλά για τα θέματα της ειρήνης και της ασφάλειας πρέπει μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι ως προς τη συνεργασία. Για το θέμα τώρα των λεπτών θεμάτων προς συζήτηση πρέπει να διαχωρίσουμε τις πολιτικές δηλώσεις από εκείνες όπου μερικοί προσπαθούν να βάλουν ε, θέσεις όπως για την Ουγκάντα, για την Ιγυρία, για την ομοφιλοφιλία, από, να το χωρίσουμε από την ποιότητα των εργασιών για τα ανθρώπινα δικαιώματα γενικά. Σας υπενθυμίζω ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο είχε αποφασίσει να δημιουργηθεί μια ομάδα εργασίας νομομαθών από τις δύο υπήρους. Υπάρχουν λοιπόν τρόποι διαλόγου και τεχνικής συνεργασίας που μπορούν να βοηθήσουν στην πρόοδο και σε μεγαλύτερο κοινό, περισσότερο κοινό διάλογο. για τους στόχους της χιλιετίας, τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας, όλοι οι συνομιλητές μας παρατήρησαν ότι η εταιρική σχέση Euh, με τα OMD ήταν προβληματική. Αλλά ότι το θέμα είναι σφαιρικό, δεν είναι συγκεκριμένο. Δεν το είπε πριν. Αρχικά. Το ECDPM επεξεργάζεται για το 2015 τι θα προβλέψει για την ανάπτυξη είναι ένα γενικότερο και πολύ πολύπλοκο πλαίσιο διαπραγμάτευσης και χρειάζεται εδώ ισορροπιστής για να τα εξισορροπήσει όλα, ακροβάτης. Το θέμα για μας όμως είναι πώς θα συνδεθεί το στρατηγικό πλαίσιο με την συγκεκριμένη εφαρμογή και αυτό θα γίνει σε επίπεδο κρατών ή εθνών και εδώ η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης είναι ουσιώδης. Αν δεχτούν όσο περισσότερο δέχονται τον κοινό προγραμματισμό τόσο πιο πολύ τόσο σαφέστερη θα είναι και η θέση τους γενικότερα για την Αφρική. Έχουμε περάσει από μία και μόνη στρατηγική για ολόκληρο τον κόσμο σε στρατηγική που καταχωρίζεται περιφερειακά όπως για το Σαχέλ και αυτό είναι ιστορική εξέλιξη και πρωτοφανής. Και αυτό το στατικό πλαίσιο ή αυτά τα στατικά πλαίσια βοηθούν την Ευρώπη και τα κράτη της να δουν τα πράγματα πιο συγκεκριμένα και ως προς τους Αφρικανούς συνομιλητές τους. Πρέπει λοιπόν να, είμαστε να έχουμε τη διανοητική τιμιότητα να αναγνωρίσουμε ότι παρά τις επικρίσεις που μπορούμε να έχουμε έχουν υπάρξει και επιτεύγματα θετικά. Γιατί είναι και πρότυπα θα αποτελέσουν αυτά. Τέλος για τον ιδιωτικό τομέα. Το CDPM έκανε μελέτες για τον ρόλο του ιδιωτικού τομέα στην ανάπτυξη σήμερα Υπάρχει το θέμα του πώς μπορούν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να συνεργαστούν με τον ιδιωτικό <laughs> τομέα και ως προς τις επενδύσεις και ως προς την οικονομική διπλωματία τους. Δηλαδή, είμαστε έτοιμοι να θεωρήσουμε ως απαραίτητο ότι πρέπει να υπάρχει μία προώθηση των ευρωπαϊκών επενδύσεων στις αφρικανικές χώρες, συλλογική προώθηση δηλαδή να έχουν ρόλο να παίξουν τα ευρωπαϊκά επιμελητήρια. Και δεύτερο ερώτημα είναι πώς θα συνεργαστούν οι οργανισμοί της βοήθειας με τον ιδιωτικό τομέα. Και αυτό είναι θέμα που έχει συζητηθεί λεπτομέρό στο ECDPM και αποσαφηνίζει τα διάφορα προγράμματα συνεργασίας που μπορούμε να εφαρμόσουμε με τον ιδιωτικό τομέα. Ευχαριστώ και με συγχωρείτε αν μακρηγόρησα κυρία Πρόεδρε μου. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε την ημερησία διάταξή μας. Ανταλλαγή απόψεων. Παρουσία του κύριου Μίχαελ Γκάλερ, ο οποίος είναι πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο και γνωρίζετε ότι κανονικά αυτή η συνεδρίαση θα πρέπει να γινόταν παρουσία του Προέδρου Μπροκ, Προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών, αλλά δεδομένης της επικαιρότητος ο κύριος Μπροκ ε, κολλείεται. Λοιπόν, προετοιμασίες της ε, κοινοβουλευτικής διάσκεψης Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής 31 Τρίτου και 1η Τετάρτου λαμβάνει η χώρα. Είναι τέταρτη σύνοδος κορυφής ε, που θα ακολουθήσει στις 2 και 3 Απριλίου την επομένη και μεθεπομένη και θα συγκεντρώσει ηγέτες από την Αφρική, την Ευρώπη, καθώς επίσης και ε, τους προέδρους των θεσμικών οργάνων Ευρωπαϊκής και Αφρικανικής Ένωσης. Η διακοινοβουλευτική διάσκεψη θα γίνει παρουσία ε, του Προέδρου Σούλτς βεβαίως και του Προέδρου Αμαντή που είναι ομόλογος του στο Παναφρικανικό Κοινοβούλιο. Θα έρθει και η κυρία Λέδη Άστον Ο Επίτροπος της Αφρικανικής Ένωσης ε, για πολιτικά ζητήματα, διάφορες υπηρεσίες και πολλές ΜΚΟ θα συμμετάσχουν. Η κοινοβουλευτική διάσκεψη θα προετοιμάσει και κοινή δήλωση που θα παρουσιάσουν οι δύο πρόεδροι του κοινοβουλίου στις 2 Απριλίου στην αρχή της 4ης Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής αυτή η διακήρυξη θα πρέπει κανονικά να συμπεριλαμβάνει τις ε, απόψεις και τα μελήματα των ε, δύο κοινοβουλίων. Ο κύριος Μιχαήλ Γκάλερ είναι πρόεδρος ε, της αντιπροσωπείας μας με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο και θα μας ενημερώσει τώρα για τις προπαρασκευαστικές εργασίες αυτής της κοινοβουλευτικής διάσκεψης. Δεν χρειάζεται να σας θυμίσω αγαπητέ κύριε Γκάλε πόσο προσφελής είναι η Αφρικανική Ήπειρος και στις δύο επιτροπές μας. Η Επιτροπή Εξωτερικών για την Εξωτερική Πολιτική και την Κοινή Ασφάλεια στην έκθεσή τη. εκφράζει τη λύπη τη για την ε, κοινή στρατηγική και ε, το γεγονός ότι έχει αποδυναμωθεί στα οχτώ σημεία της, ε, γιατί υπάρχουν περιτές ε, συμφωνίες ε, με διάφορους εταίρους που επικαλύπτονται, ενώ λείπουν τα απαραίτητα κονδύλια. Τονίζει η Επιτροπή Εξωτερικών ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε πέρα από το απλό θέμα του capacity building, της ε, οικοδόμησης ικανοτήτων και να έχουμε στόχο μια πραγματική εταιρική σχέση για την ασφάλεια, τη συνεργασία, την ειρήνη και με τις περιφερειακές οικονομικές συνεργασίες για να έχουμε μια ουσιαστική ευρωαφρικανική εταιρική σχέση. Αγαπητέ κύριε Γκάλερ, ως πρόεδρος της αντιπροσωπείας μας, λοιπόν, θα σας παρακαλούσα να μας πείτε τι προτίθεστε να κάνετε για να εκφράσετε τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις επαφές που έχετε με τους Αφρικανούς ομολόγους σας και τι περιμένετε γενικότερα από αυτή την τέταρτη σύνοδο κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής. Θα σας ακούσουμε πολύ προσεκτικά, ιδιαίτερα για τον τρόπο με τον οποίο η κοινή κοινοβουλευτική ε, διακήρυξη θα μπορούσε να ενισχύσει το ρόλο των κοινοβουλίων στην κάθε Ήπειρο για να λογοδοτούν οι, ε, για την πολιτική ασφαλείας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην Αφρική και να μπορούν όλοι οι πολίτες και των δύο υπήρων να ε, είναι ενήμεροι για τα αποτελέσματα αυτών των πολιτικών. La discussion politique... Η πολιτική συζήτηση θα γίνει κατά τη διάρκεια της ίδιας Συνόδου Κορυφής και θα πρέπει από τώρα να σκεφτούμε τι ρόλο θα διαπαθαρματίσει και στην κοινοβουλευτική διάσκεψη για να δούμε πώς εμείς θα ε, κάνουμε αυτές τις σκέψεις μας να αντανακλώνται στα τελικά κείμενα μετά τη Σύνοδο. Παρακαλώ κύριε Γκάλερ, έχω τη χαρά να σας δώσω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, και εγώ θα επιθυμούσα να ε, γίνει η συνεδρίαση αυτή κοινή με την Επιτροπή Εξωτερικών όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί και σε μεγαλύτερο πλαίσιο και ευρύτερο με τις διεπιτροπές, αλλά όπως είπατε πρόεδρε, η επικαιρότητα και οι εξελίξεις στην Ουκρανία μας έχουν ξεπεράσει και αυτό το χρόνο χρειάστηκε η Επιτροπή Εξωτερικών να το διαθέσει τον Μπόρι Τάρασιουκ που είναι ο Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ουκρανίας και αυτή τη στιγμή είναι στην Επιτροπή ε, ΑΦΕΤ. Και επειδή και εγώ εμπλέκομαι πολύ στα θέματα της Ουκρανίας ήμουν απόν στην προηγούμενη παρουσίαση γιατί ε, ε, άκουσα τα όσα είχαν να μας πούν για τα τεκτενόμενα στην Ουκρανία. Παρ' όλα αυτά έχω πάρει έγγραφα στα αγγλικά, έχω προετοιμάσει στα αγγλικά και θα τα πω και στα αγγλικά. Αγαπητοί συνάδελφοι, γνωρίζετε ότι η πρώτη σύνοδος κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής ήδη έλαβε χώρα στο Κάιρο το 2000. Ε, μόλις όμως τη δεύτερη σύνοδο κορυφής, τη Λισαβόνα το Δεκέμβριο του 2007, ε, πήρε την ε, σωστή μορφή αυτή η σύνοδος και λήφθη η απόφαση ανατριετία να διοργανώνονται Συνεδριάσει ε, τη μια φορά στην Αφρική, την επόμενη στην Ευρώπη. Και τότε εγκρίθηκε και η διακήρυξη της Λισαβόνα. Η κοινή στρατηγική έχει ε, ως περίγραμμα ένα όραμα για μια μακροπρόθεσμη στρατηγική και συνεργασία μας σε ένα παγκοσμιωμένο κόσμο. Πέρα από την αναπτυξιακή συνεργασία έχουμε και θέματα κοινού πολιτικού ενδιαφέροντος. Πέρα από την Αφρική και προετοιμάζουμε και το έδαφος για γενικότερα ζητήματα και παγκόσμια και ευρωπαϊκά, όχι μόνο αφρικανικά. Ξεπερνάμε τον κατακαιρματισμό και υποστηρίζουμε την Αφρική ε, στην ε, αγωνία της να βρει και περιφερειακές και υπηρετικές λύσεις για τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Βεβαίως με θεσμούς για καλύτερη συμμετοχή των πολιτών και των Αφρικανών και των Ευρωπαίων για να ενισχυθεί η κοινωνία των πολιτών στις δύο υπήρους. Έχουμε κοινό όραμα και κοινέ αρχές άλλωστε. Και έτσι ορίζεται και η στρατηγική σε 8 ειδικέ σχέσει. Η τρίτη σύνοδος έγινε στην Τρίπολη τον Νοέμβριο του 2010 με μια διακήρυξη και ένα δεύτερο πρόγραμμα δράσης. The fourth summit between the 54 states of the... Και είναι 54 τα κράτη, ξέρετε, της Αφρικανικής Ένωσης και 28 βεβαίως της ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και 2 και 3 Απριλίου θα είναι η επόμενη σύνοδο. Δεν είναι Αφρικανική Ένωση αυτό, αλλά ε, με έναν τρόπο που να μπορέσει να συμμετέχει και το Μαρόκο ένα σχήμα. Ε, προηγείται, όπως είπατε, κοινοβουλευτική διάσκεψη που για πρώτη φορά επίσης διοργανώθηκε στη Λισαβόνα το 2007. Παραμονές ε, Τη δεύτερη και στη συνέχεια στην Τρίπολη τη Τρίτη. Εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα γίνει αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 31 Μαρτίου και 1 Απριλίου. Πέρσι τον Οκτώβριο για την προσωπία μας είχαμε μια κοινοβουλευτική συνεδρίαση με ε, του συναδέλφους στη Νότιο Αφρική στην έδρα του Κοινοβουλίου για να προετοιμάσουμε τη συνεδρίαση αυτή. Και θεωρήθηκε ότι έχει εδρεωθεί πλέον και καθιερωθεί αυτή η πρακτική να προηγείται κάθε φορά τη Συνόδου Κορυφής μια κοινοβουλευτική διάσκεψη. Συμφωνήθηκε και η μερίσια διάταξη μεταξύ άλλων και το σχήμα να γίνεται ακριβώς στις παραμονές της Συνόδου Κορυφής να έχει διάρκεια τριών μισών ημερών, αρχίζει δηλαδή το πρωί, ε, τώρα προκειμένου στις 31 Μαρτίου και ένα κοινό σχέδιο, σχέδιο κοινή δήλωση μάλλον θα προετοιμάζεται βάσει των εκτιμήσεων των στρατηγικών. Η κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να συμμετέχει και οι ε, ενεχόμενες μη κυβερνητικές οργανώσεις να ενημερώνουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Αφρικανικό στο περιθώριο όλων αυτών των συναντήσεων. Το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων των μονίμων αντιπροσωπιών για το πρώτο ήμιση του 2014 έχει εγκριθεί από τη διάσκεψη των Προέδρων στις 12 Δεκεμβρίου του 2013 και συμπεριλαμβάνει και αυτό την προσύνοδο, για να την πω έτσι. Για τη συμμετοχή γνωρίζετε ότι το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο θα εκπροσωπηθεί από 23 ε, μέλη και μια ad hoc αντιπροσωπεία θα έρθει απέναντι ε, ε, ισομερής 23 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από τους 23 ο ένας θα είναι ο πρόεδρος Σούλτς και 12 τα μέλη της αντιπροσωπείας και οι υπόλοιπε 10 θέσεις θα μοιραστούν σύμφωνα με τις πολιτικές ομάδες και κυρίως μέλη της ΑΦΕΤ, ΔΕΒΕ, ΙΝΤΑ και ε, της ΑΚΕ. Να σας πω ειλικρινά, ελπίζω και πιστεύω να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε 23 άτομα και να μην ψάχνω να κοιτάω από ποια θεσμικά όργανα καθένας από, ε, ε, από ποια ε, επιτροπή, αντιπροσωπεία. Αν μετρήσουμε όλα τα πλήρη και τα πραγματικά μέλη, νομίζω θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε 23 άτομα, όχι μόνο για τα εγγένεια, αλλά και για καθ' τη διάρκεια και τις τρεις μισές ημέρες να είμαστε παρόντες και να συζητήσουμε θέματα ενδιαφέροντος με τους Αφρικανούς συναδέλφους και να μην δώσουμε κακή εικόνα. Γνωρίζω ότι πολλοί από εμά είμαστε σε προεκλογική εκστρατεία και όλα αυτά τα ζητήματα που μας απασχολούν παραμονές εκλογών είναι γνωστά. Αλλά παρακαλώ έκκληση προς όλους να έχουμε μια παρουσία έτσι που να μην μας εκθέσει. Στις 12 Μαρτίου θα συνεδριάσουν αυτά τα 23 μέλη στο Στρασβούργο για να συγκροτηθούν σε σώμα. Ένα σχέδιο ε, τεχνικό της κοινή διακήρυξης θα έχει προετοιμαστεί και θα συμπεριλάβουν και τη μελέτη που μόλις παρουσιάστηκε, τα έγγραφα αυτά, της ECDPM για την εφαρμογή της κοινή στρατηγικής Αφρικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ε, είναι πολύτιμη η συνεισφορά όλων των μελών και για τα 23 μέλη. Ξέρουμε ότι η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΑΕΔ είναι να περιορίσουν τον αριθμό προτεραιοτήτων την επόμενη τριετία, να εστιάσουν σε λίγους τομείς που μπορούν να δώσουν καλά αποτελέσματα. Δεν λέω να το σεβαστούμε απολύτω, αλλά το σκεφτούμε κι εμεί. Μήπω χρειάζεται περιορισμό στον αριθμό των προτεραιοτήτων. Προσωπικά θα πρότεινα να επικεντρωθούμε στα εξή να συνεχίσουμε τα όσα έχουμε ήδη επιτύχει στην ασφάλεια και την ειρήνη. Είναι από τα θέματα που είχαν τα πιο απτά αποτελέσματα. Δεύτερο. Ενίσχυση μακροοικονομικής συνεργασίας στα πλαίσια της δημογραφικής εξέλιξης και του νέου δυναμισμού, όπως τον αντιλαμβάνεται η Αφρική, θα πρέπει να δημιουργηθούν θέσει απασχόληση. Έτσι λοιπόν πρέπει να υποστηριχθούν αυτές οι δράσεις. Τώρα, για τα βήματα και τις κινήσεις που θα γίνουν υπηρετικά ώστε να μπορέσουν τα εθνικά συστήματα ασφάλισης ε, να αναπτυχθούν. Ένα πιλωτικό πρόγραμμα πρέπει να εκπονηθεί με βάση τις ε, βέλτιστες τεχνολογίες όσον αφορά την ε, υγιεινή των τροφίμων, του νερού και τις κλιματικές αλλαγές. Το πρόγραμμα θα πρέπει να δούμε ότι θα πρέπει να έχει ως εξής. Δευτέρα πρωί ε, ματιού έναρξη με προσφώνηση του Πρόεδρου Σούλτς και του κυρίου Αμαντή Κάθριν Άστον και Αΐσα Αμπτουλάχη. Ε, ε, Αφρικαν, Αφρικανός Επίτροπος ε, για αυτά τα θέματα. Θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων το απόγευμα μεταξύ ΜΚΟ και Κοινωνίας των Πολιτών. Θα συνεχίσουμε με την πρώτη συντακτική συνέλευση για μια κοινή διακήρυξη. Τρίτη πρωί θα αρχίσει η συζήτηση για τα θέματα δικαιωμάτων του ανθρώπου για μια κοινή στρατηγική. Θα ακολουθηθεί από τα τελικά σχόλια και την κοινή διακήρυξη και έγκρισή της. Θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα στο επίπεδο μιας όπου θα συμμετάσχει στην Κοινοβουλευτική Σύνοδο Κορυφής. Έχουμε, πιστεύω με αυτόν τον τρόπο, πολλές ευκαιρίες, ευρύτερες ευκαιρίες, ώστε πηγαίνοντας προς αυτή την συνάντηση μέχρι τα τέλη Μαρτίου να εξετάσουμε ποιες θα είναι οι προτάσεις από πλευρά συναδέλφων και ποια μορφή θα πάρουν. Από πλευρά της αντιπροσωπείας μας έχουμε μια και εργάστηκαν για ένα σχέδιο εγγράφου και θα είναι κάτι κοινό όπως επιθυμούμε το αποστήλαμε αυτό το ε, προκαταρκτικό σχέδιο τους συναδέλφους, συναδέλφους μας και ζητήσαμε να υποβληθούν σχόλια από πλευράς τους πριν από την επίσημη ας εμπλοκή των ε, συναδέλφων εδώ. Είμαι όμως βέβαιος ότι οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι ήδη έχουν ε, δει αυτό το προκατακτικό προσχέδιο προτού επίσημα υποβληθεί στη συνέχεια στις διαβουλεύσεις προς έγκριση και ενταχθεί ε, και εγκριθεί από πλευράς μας. Αυτό γενικά από εμάς κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους είναι κάτι που σε σχέση με τις συνεδριάσεις μας ε, έχουμε την εντύπωση ότι η πολιτική δέσμευση από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφέρω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ε, ή τη μία ή την άλλη κατά πρώτο λόγο δεν υπάρχει άμεση εμπλοκή επιτόπου. Η πολιτική λοιπόν φιλοδοξία να μπορέσει να λειτουργήσει αυτή η συνεργασία Ευρώπης-Αφρικής ως μια προτεραιότητα δεν έχει ακόμα φτάσει στα αναγκαία επίπεδα από πλευράς μας και κυρίως δεν έχουν υπάρξει τακτές ε, υπουργικές ε, συναντήσεις ε, και για τις δύο επιτροπές ναι δεν έχουν συναντηθεί αλλά στο επίπεδο της εξωτερικής υπηρεσίας δράσης δεν είχαμε ακόμα υπουργικές τριμερείς και ασκήσαμε, διατυπώσαμε παράπονα εδώ και πολύ χρονικό διάστημα ότι από και από πλευράς των Αφρικανών έχει αυτό διατυπωθεί ως, ως παράπονο ότι δηλαδή δεν τα παίρνουμε τα πράγματα όσο σοβαρά όσο θα έπρεπε και δεν έχει επιτευχθεί εκείνο το οποίο θα μπορούσε να είχε επιτευχθεί από πλευρά μας στα διαφορετικά αυτά θέματα. Αυτή η επίκριση λοιπόν για την αντιμετώπιση της οποίας την χάνει με την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για τα θέματα της Αφρικής είναι κάτι το οποίο εμφαίνεται όχι μόνο στα έγγραφα αυτά αλλά αντανακλάται και ε, βρίσκει απήχηση και στις συζητήσεις μας και πρέπει να δούμε πώς θα ανταποκριθούμε και πώς θα καταφέρουμε στο μέλλον να είμαστε πιο αποτελεσματικοί να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε μια άλλη τάση και πορεία. Δεν είναι μόνο το θέμα των ατόμων που εμπλέκονται, αλλά είναι και το θέμα των ζητημάτων, των θεμάτων. Ποια προτεραιότητα τους δίνουμε και πώς τα προάγουμε συγκεκριμένα. Αυτό θα είναι ένα θέμα το οποίο έχει ύψιστη προτεραιότητα. Ολοκληρώνω εδώ και θα ακούσω τις παρατηρήσεις των συναδέλφων. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Μαρτίνες. Ευχαριστώ Μιχαήλ. Γκάλερ. Ευχαριστώ πολύ. Προτού καταλήξουμε σε αυτό το θέμα, σε σχέση και με την παρουσίαση κιόλας ε, για την έκθεση, ενδιαφέρουσα παρουσίαση που μας παρουσιάστηκε πιο πριν από τον κύριο Έλλη που είχαμε, υπήρξαν κάποια σχόλια επί κάποιων πραγμάτων. Εγώ θα ήθελα μόνο να σου θέσω δύο ζητήματα, δύο θέματα που πιστεύω ότι δεν μπορούν να απουσιάζουν, δεν μπορούν να αμεληθούν σε αυτό το πλαίσιο. Ένα από αυτά τα θέματα. Είδα ότι υπάρχει ένας χώρος που προβλέπεται για το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πιστεύω ότι μέσα στο πλαίσιο των δικαιωμάτων του ανθρώπου θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο το θέμα της νομοθεσίας και των διατάξεων όχι ομοφοβικών αλλά θα έλεγα καταδίωξης και διωγμού της ομοφιλοφιλίας. Κατά κάποιο τρόπο δηλαδή μια επιδίνωση και οπισθοδρόμηση ως φαινόμενο. Και το βλέπουμε αυτό και στην Ουγκάντα, αλλά και σε άλλες χώρες. Στην Ιγυρία για παράδειγμα που είναι μία από αυτές τις χώρες όπου και αυτό αναφύεται, παρουσιάζεται ως φαινόμενο. Δεν θα είναι δυνατό να αποφύγουμε λοιπόν πιστεύω μια συζήτηση για αυτό το θέμα. Και θα είναι σίγουρα ένα περίπλοκο θέμα. Υπάρχει όμως ένα άλλο θέμα το οποίο δεν αναφέρθηκε εδώ καθόλου και το οποίο πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ θεμελιώδους σημασίας, πολύ σημαντικό. Με ανησυχεί ότι ακούμε κάθε μέρα να γίνεται λόγος για το boom, για την έκρηξη αυτή στην Αφρική, όμως για να δούμε, συνεχίζει να υπάρχει να, υπάρχει πάνω από, να υπάρχουν πάνω από 50.000 υποσαχάριοι πολίτες που περιμένουν σε ένα δάσος ε, στο Μαρόκο για να περάσουν το φράχτη και να περάσουν στην Ευρώπη, δηλαδή στη Θέουτα και Μελίγια, για να μπορέσουν να περάσουν μετά στην Ισπανία. Παίζουν κορώνα γράμματα τη ζωή τους, παίζουν τη ζωή τους θα έλεγα ρίχνοντας αυτή τη ζαριά προσπαθώντας να περάσουν το φράχτη. Και εδώ πάλι υπάρχουν, κάτι, το, υπάρχουν πράγματα τα οποία πολλοί Ευρωπαίοι αγνοούν ή περιφρονούν. Και έχουμε εδώ και μια συνάντηση των Υπουργών, ε, ε, των Εσωτερικών και υπάρχει και ο Υπουργό Εσωτερικών της Ισπανίας ε, για να συζητήσει με την κυρία Μάλστρομ για αυτά τα θέματα. Έχουμε συζητήσει πάρα πολύ για τη Λαμπεντούζα της Ιταλίας, αλλά γίνεται και συζήτηση για το, αυτό που συμβαίνει σε μια ολόκληρη σειρά ε, ε, πολιτών της Αφρικής από την Μεσημβρινή Αφρική, από την Υποσαχάρια Αφρική που ε, προσπαθούν να εισέλθουν στην Ισπανική επικράτεια και τους πυροβολούν με σφαίρες, λαστιχένιες σφαίρες και είχαμε και 15 νεκρούς εκεί. 15 βέβαια είναι τα πτώματα τα οποία συνελέγησαν. Δεν ξέρουμε πόσα είναι τα πτώματα τα οποία δεν έχουν συλλεγεί και πόσα είναι τα θύματα. Κάνουμε λόγο για μια πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση. Και θα είναι λοιπόν λοιπόν πραγματικά συγχώρητο σε αυτή τη σύνοδο Κορυφή το θέμα της μετανάστευσης να μην είναι ένα θέμα το οποίο να έχει πραγματικά ένα πριτανεύοντα κυρίαρχο ρόλο στις συζητήσεις και έναντι των εταίρων μας στην Αφρική, των Αφρικανών εταίρων πρέπει να θέσουμε στο τραπέζι ποια είναι η κατάσταση και να δούμε πώς βλέπουν και αξιολογούν εκείνη μια κατάσταση που πραγματικά είναι πολύ προβληματική και που πραγματικά ε, πρέπει να πούμε ότι ε, ξεπέρασε πλέον τα όρια και έχει φτάσει σε μια κατάσταση που πρέπει να βρούμε λύσεις ε, για αυτήν και για την κοινωνικο οικονομική κατάσταση σε αυτές τις χώρες και τους Αφρικανούς που αναγκάζονται να φύγουν από εκεί για να έρθουν στην Ευρώπη αλλά και όλα τα προβλήματα που συνεπάγεται αυτό για την Ευρώπη και την κατάσταση που δημιουργεί για αυτήν. Αυτή είναι η πρόθεσή μας λοιπόν. Να συζητηθεί αυτό σε αυτή τη σύνοδο όπως και στη Λισαβόνα και στην Τρίπολη και θα συνεργαστούμε μαζί σου να κάνουμε ό,τι χρειάζεται ώστε αυτή η συνεδρίαση να είναι επικοδομητική και να είναι μια καρποφόρα συνεδρίαση που θα δώσει αποτελέσματα και να έχει έχει και χειροπιαστές ε, επιπτώσεις και για τη διακυβερνητική αυτή ε, διάσκεψη έχει πολύ μεγάλη σπουδαιότητα αυτό. Ευχαριστώ. Merci Je donne Ευχαριστώ πολύ. Η Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων, ο κύριος Ντοκώστα Περέρα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και κύριε Μιχαήλ Γκάλερ για όλες τις πληροφορίες που μας δώσατε για τη διάσκεψη που νομίζουμε ότι θα είναι πολύ καλή ευκαιρία για το Παναφρικανικό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να συζητήσουν τις σχέσεις τους. Είναι μια ευκαιρία που μας ενδιαφέρει και μας πολύ. Απλώς λυπούμαστε γιατί δεν κατέστη δυνατόν να συναντηθούν πιο νωρίς οι βουλευτές μεταξύ τους. Τέλος πάντων, αναμένουμε ο πρόεδρος Σούλτς να μπορέσει να λάβει το λόγο στη διάσκεψη ώστε να ακουστούν και οι δικές σας ανησυχίες. Πολύ λογικό θα ήταν να συνδυάσουμε τις δικές σας ανησυχίες και ενδιαφέροντα με εκείνα τους διάσκεψης γιατί η ειρήνη και η ασφάλεια φυσικά είναι από τα πιο σημαντικά θέματα της διάσκεψης καθώς και η βιώσιμη ανάπτυξη και η απασουχόληση καθώς και τα θέματα της παιδείας, capacity building, μετανάστευση. Να σας πω μερικά για τα θέματα που μας ενδιαφέρουν εμάς και το πρόγραμμα των συζητήσεων. Δηλαδή, φυσικά θα υπάρξουν λόγοι και συζητήσεις. Ακόμη πιο σπουδαίο όμως είναι τι θα αφήσει η διάσκεψη ως κληρονομιά, γραπτά έγγραφα, έγγραφα δηλαδή, πέραν των πολιτικών δηλώσεων που γίνονται συνήθως σε όλες τις διασκέψεις. προτίθεται να υπάρξει ένα προγραμματικό κείμενο που να συνοψίζει από ποσοτικής απόψεως ποια ήταν η σχέση μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής από το 2007, οπότε εγκρίθηκε η πρώτη κοινή στρατηγική. Επίσης συζητούμε με τους Αφρικανούς συνομιλητές μας τη δυνατότητα στις πολιτικές δηλώσεις να προσθεθούν μερικά συγκεκριμένα μερικές συγκεκριμένες λεπτομέρειες όπου ελπίζουμε να υπάρξει σημαντική πρόοδος. Τέσσερα σημεία δηλαδή κυρίως που θέλουμε να συζητήσουμε με την αφρικανική πλευρά και είναι οι κλιματολογικές αλλαγές, η γεωργία, η μετανάστευση και η περίοδος μετά το 2015 Μπορώ να σας πω ήδη ότι και τα τέσσερα αυτά θέματα θα συζητηθούν και γραπτός στα έγγραφα της διάσκεψης. Θέλουμε όμως να έχουν νόημα όλα αυτά. Αν δεν έχουν νόημα καλύτερα να μην υπάρξουν. Είτε να γραφτεί κάτι καινούριο και ουσιώδες, έστω και μία-δύο παράγραφοι στη Γενική Δήλωση για που να δείχνει πού υπάρχει η συμφωνία μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής. Ελπίζουμε λοιπόν να έχουμε ένα αποτέλεσμα θετικό και για τις δύο πλευρές ώστε οι δηλώσει να συμπεριληφθούν γραπτός στα αποτελέσματα της διάσκεψης. Επειδή πρόκειται για σχέση μεταξύ ίσων, θέλουμε η καταπολέμηση της ανέχειας στην Αφρική να μην αφορά μόνο τη χορήγηση βοηθείας αλλά και τις επενδύσεις και το εμπόριο. Ε, αυτό θέλουμε να τονιστεί στη Σύνοδο. Η ιδέα σας λοιπόν για την ενίσχυση της <coughs> ειρήνης και της ασφάλειας της μακροοικονομικής διακυβέρνησης της απασχόλησης της χρήσης των καλύτερων δυνατών τεχνολογιών θα τέριαζε πάρα πολύ καλά και με τις δικές μας ιδέες και μπορούμε να τα συνδυάσουμε όλα αυτά. Τώρα, ποιο θα είναι το σύστημα ασφαλείας δεν το ξέρω, θα είναι κάτι πιο δύσκολο σίγουρα, αλλά οποιαδήποτε ιδέα προέλθει από το Κοινοβούλιο θα γίνει δεκτή με τη δέουσα προσοχή από εμά. Βέβαια κάθε πολιτική δήλωση είναι συμβιβασμός. γιατί θα περάσει μόνο ότι είναι αποδεκτό και από τις δύο πλευρές. Μπορούμε να αναμένουμε λοιπόν δύσκολες διαπραγματεύσεις και τα αποτελέσματα δεν θα είναι ούτε αυτό που θέλαμε εμείς, ούτε αυτό που ήθελαν οι Αφρικανοί, αλλά θα μπορέσουμε ίσως να τα γεφυρώσουμε. Γιατί πρόκειται για δύσκολα προβλήματα στις σχέσεις μας και αναμένω ότι θα υπάρξει ελεύθερη συζήτηση στη διάσκεψη και ότι δεν θα υπάρξουν ταμπού ή φόβοι. Ξέρουμε ότι έχουμε διαφωνίες για μερικά θέματα, αλλά θα συζητηθούν και αυτά. Ίσως να μην φαίνονται οι συζητήσεις και οι διαμάχες αυτές στην πολιτική δήλωση, αλλά θα θέλαμε το κοινό να μάθει τουλάχιστον τις ιδέες όπου συμφωνούμε και όπου μπορεί να υπάρξει πρόοδος. Θα ήταν πολύ βοηθητικό να υπάρξει μια Δήλωση που να λέει αυτά λένε οι Αφρικανοί, δεν θα ήταν πολύ βοηθητικό αν λέγαμε οι Αφρικανοί λένε το α και οι Ευρωπαίοι το μείον α. Θα θέλαμε λοιπόν την κατανόησή σας για τις δυσκολίες επίτευξης ενός κοινού κειμένου που δεν σημαίνει ότι ούτε θα αποτεφευχθεί ούτε θα συζητηθεί κατά ανάγκη όλο το δύσκολο θέμα, όποια δύσκολο θέμα υπάρχει και σας εύχομαι καλή επιτυχία και προσβλέπουμε και εμείς στα συμπεράσματα της διάσκεψής σας ελπίζοντας να παίξουμε και εμείς κάποιο ρόλο. Ευχαριστώ. Merci beaucoup. Ευχαριστώ πολύ. Θα ξαναδώσω το λόγο στον κύριο Γκάλερ για να ολοκληρώσει. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να επικεντρωθώ στο εξή σημείο καταρχάς. Νομίζω ότι θα έχουμε εκτενέστατες συζητήσεις για το θέμα των ε, προσφύγων και της μετανάστευσης. Και ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγματικά θα πρέπει να διατρανώσουμε ότι δεν επιτρέπεται το εξή. Πέρα από το γεγονός ε, ότι τελικά τις πρόσφυγες τους υποδεχόμαστε. ότι δεν μπορούμε να επιτρέπουμε να πεθαίνει ο κόσμος ερχόμενο στην Ευρώπη, είτε από δική μας δράση, δηλαδή να τους πυροβολούμε, είτε από δική μας αδράνεια να τους αφήνουμε να πνίγονται. Αυτό δεν επιτρέπεται. Θα πρέπει να το συζητήσουμε φιλικά με τους Αφρικανούς, αλλά να, δεν επιτρέπεται ο κόσμος που θέλει να έρχεται στην Ευρώπη να πεθαίνει στο δρόμο. Αυτό είναι μια πολιτική αξίωση που θα πρέπει να διατρανώσουμε. Από εκεί και πέρα βλέπουμε τι, τι κάνουμε. ποιο μπορεί να παραμείνει και ποιο δεν μπορεί. Αυτό είναι τελείω διαφορετικό θέμα. Αλλά το πρώτο βήμα είναι κάτι που εξαρτάται από τις δικές μας πράξεις και παραλήψεις, αλλά δεν επιτρέπεται να αφήνουμε τους ανθρώπους να πεθαίνουν. Αλλιώς δεν μπορούμε να συζητήσουμε για άλλες πολιτικές με την Αφρική. Μειώνοντας τα θέματα θα εστιάσουμε καλύτερα και θα θα συγκεκριμενοποιήσουμε και θα έχουμε και απτή χειροπιαστή πρόοδο και ως Κοινοβούλιο. Το σημειώνουμε αυτό. Και ελπίζω πάρα πολύ και τους συθήνοντες στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης να τα πείτε αυτά και στους υπουργούς να επαναληφθεί ο τακτικός πολιτικός διάλογος μετά από τις Σύνοδο Έχουμε σε επίπεδο υπουργών τρόικες και το είχαμε παγίως εδώ και καιρό. Δηλαδή, κάθε φορά πριν συνεδριάσουν αυτοί οι τρεις υπουργοί, ε, είχαμε και μια επαφή με την κοινοβουλευτική διάσταση, ας πούμε σε ένα ε, πρόγευμα εργασίας, με κάποιο τρόπο να έχουμε και την κοινοβουλευτική μας παρουσία. Αλλά επειδή είχαν καταργηθεί αυτέ οι συνεδριάσεις δεν μπορούσαμε εμεί ως κοινοβούλια να πούμε τη γνώμη μα. Έχουμε και πολύ μεγάλο ίδιο συμφέρον, αν θέλετε, γιατί το είχαμε συμφωνήσει να εχουμε τέτοιε επαφέ επαφές back-to-back meetings. Θα πρέπει να πιέσει και η κυρία Άστον και ο κύριος Φανρομπόη και ο κύριος Μπαρόζο και οι τρεις τους ε, και από πλευρά μα, εμεί, στη Σύνοδο Κορυφή, να συγκεντρώσουμε του πρωθυπουργού, του ηγέτε, όχι μόνο υπουργού εξωτερικών ή υπουργού αναπτυξιακή βοήθεια ή κανέναν υφυπουργό να στείλουν. Ε. Νομίζω ότι έχουμε και την πολιτική αξίωση αυτή τη σύνοδο κορυφή να είναι κορυφή Και από τους 28 να μην λείπει κανείς και σε επίπεδο πρωθυπουργού μάλιστα. Αυτό θα μπορούσαμε να το διαβιβάσουμε και ως μήνυμα σε σχέση με όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Merci beaucoup. Ε, και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Γκάλε και όλους ε, σας. Θα κάνουμε μια διακοπή τώρα μέχρι τις 5 παρα 10 για να συνεχίσουμε ε, με την ανταλλαγή υπόψη με τη Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ για να συζητήσουμε τις ανθρωπιστικές κρίσεις που πλήττουν την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, τη Συρία και τον Νότιο Σουδάν. Μικρή διακοπή 10 λεπτών.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

Ευχαριστώ. Notre séance reprend. Je souhaite la bienvenue au directeur général de la M. Klaus. Επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση. Καλωσορίζω τον κύριο Σέρενσεν. Έξι εβδομάδες πριν σας είχαμε ακούσει για τις κρίσεις στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, στη Συρία και τον Νότιο Σουδάν. Δυστυχώς αυτό το τελευταίο διάστημα δεν ε, σταμάτησε η βία σε καμία από τις τρεις χώρες και αυτό και σήμερα ερχόμαστε να το ξανασυζητήσουμε. Στη Συρία ε, δεν γνωρίζει καμία ε, ανάπαυλα η κρίση και χωρίς προοπτική για πολιτική λύση, ενώ εκατομμύρια Σύριοι χρειάζονται κατεπηγόντως ανθρωπιστική βοήθεια. Στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία περίπου ένα εκατομμύριο πολιτών φεύγουν, για να ξεφύγουν από τη βία που έχει γίνει πλέον και θρησκευτική και ανθρωπιστική κατάσταση είναι πάρα πολύ επισφαλή και για του βοηθούς εκεί στην ανθρωπιστική βοήθεια. Στο δε νότιο Σουδάν κινδυνεύει να επιδεινωθεί η κατάσταση εάν οι γεωργικέ δραστηριότητε δεν χρηματοδοτούνται τώρα που είναι η περίοδος σποράς. Θα θέλαμε να μας πείτε πώς το ανθρωπιστικό γραφείο αντιμετωπίζει ταυτόχρονα αυτές τις κρίσεις και τι αντίκτυπο μπορεί αυτό να έχει στον ε, προϋπολογισμό της Ένωσης για τα ανθρωπιστικά θέματα για το υπόλοιπο του έτους. Σας δίνω μέσα στο λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. έβα δηλαδή. Και εγώ χαίρομαι που έρχομαι να σας δω για να μιλήσουμε για μερικά θέματα στις τρεις χώρες που αναφέρατε για τις τρεις χώρες που αναφέρατε αλλά δεν μπορώ να μην μιλήσω και για την Ουκρανία Ίσως μάλιστα να αρχίσω από αυτό. Παρακολουθούμε από κοντά την κατάσταση προς το παρόν. Δεν υπάρχει ακόμη σοβαρή ανθρωπιστική κρίση. Υπήρξαν ορισμένα υγειονομικά προβλήματα, με ιατρικά προβλήματα, αλλά δεν είναι ότι δεν το σκεφτόμαστε οι διάφορα σενάρια, αλλά μπορούμε νομίζω να πούμε ότι η ανθρωπιστική πρέπει να είναι έτοιμη. Ελπίζω να μην γίνει τίποτα σοβαρό, αλλά από αυτά που βλέπουμε, αυτά που βλέπουμε είναι πολύ σοβαρά. Να ξέρετε λοιπόν ότι παρακολουθούμε τα πράγματα. Ίσως τώρα να τα πω στη γλώσσα του Νίξον, γιατί έτσι τα έχω γραμμένα. Και Καταρχήν θα ήθελα να αποτίσω ένα φόρο τιμή στην Επιτροπή σας και στον κύριο Στρίφλερ για όλα όσα έκανε για το Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών. Χάρηκα πολύ που με τέτοια πλειοψηφία εγκρίθηκε αυτό το νομοθέτημα της προάλλες στο Στρασβούργο. Και πιστεύω ότι αν και δεν θα εφαρμοστεί αμέσως, τα επόμενα χρόνια θα βλέπουμε όλο και περισσότερους νέους και λιγότερο νέους Ευρωπαίους που εθελοντικά θα βοηθούν και ελπίζω έτσι να βρούμε προσωπικό και για όλες τις ανθρωπιστικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται. Χαίρομαι λοιπόν πολύ που μπόρεσε να εγκριθεί αυτό το νομοθέτημα σε αυτήν τη θητεία ήδη. Θα ήταν σκανδαλώδες αν δεν το είχαμε καταφέρει, αλλά το καταφέραμε. Ο κυρία Στρίφλερ, εσάς ευχαριστούσα μεταξύ άλλων για όσα κάνατε για τους εθελοντάς. Χαίρομαι ιδιαίτερα για την μεγάλη πλειοψηφία που επετέχθη στο Στρασβούργο. Νομίζω ότι έτσι έχουμε ένα πολύ καλό μέσο ή εργαλείο για να κάνουμε τη δουλειά μας. Σε περιφέρειες κρίσης ιδίως. Λοιπόν, για τη Συρία τώρα. Είναι δύσκολο να υπάρχουν καλά νέα από εκεί. Να μην με παραξηγήσετε λοιπόν, αλλά θα αναφέρω μερικά στοιχεία που δεν είναι μεν καλές ειδήσει, αλλά τουλάχιστον είναι λιγότερο αρνητικές. Πρώτον, υπενθυμίζω και ευχαριστώ και σας και πολλές χώρες μέλη που τόσο στεναρά εμπνεπλάκησαν στο Κουβέιτ 2. Είναι καταπληκτικό ότι η Ένωση ολόκληρη, όλοι μαζί, χώρες μέλη, με τη στήριξή σας, η Κομισιόν, από την αρχή της διένεξης, κατάφερε να δοθούν 2,6 δισεκατομμύρια από την αρχή της σύραξης. Και η διάσκεψη Κουβέιτ 2, τα κράτη-μέλη και η Ένωση ως τέτοια, πρόσθεσαν άλλο ένα δισεκατομμύριο σε αυτά. Άρα δεν έχουμε προδώσει την θέληση των πολιτών να επιδείξουν αλληλεγγύη. Και γι' αυτό είναι καθήκον μας να διασφαλίσουμε ότι η βοήθεια πράγματι θα φτάσει σε εκείνους που τη χρειάζονται. Εκεί έχουμε πολλές δυσκολίες. Σας το έχω ξαναπεί νομίζω και άλλη φορά. Έχουμε ακόμη προβλήματα με τις θεωρήσεις, σταματάνε τα φορτηγά, τα ξεφορτώνουν, τα ξαναφορτώνουν Έχουμε τις πολιορκημένες περιοχές και άλλες που ελέγχονται από την κυβέρνηση δύσκολη κατάσταση εκεί, αλλά και περιοχές όπου ελέγχονται από τους επαναστάτες και πρέπει να γίνονται διαπραγματεύσεις και όλο πιο περίπλοκα είναι τα πράγματα. Αν υπάρχει κάποιο καλό μαντάτο έστω, θα έλεγα ότι είναι ότι επιτέλους στα Ηνωμένα Έθνη καταφέραμε να έχουμε ένα ψήφισμα για τα ανθρωπιστικά, για την ανθρωπιστική πτυχή, για την ανθρωπιστική δράση. Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε, θα μπορούσε να είναι πιο ε, ενδυναμωμένο, να υπήρχε μια παράγραφος ε, που να ε, οδηγούσε στο να ληφθούν κάποια μέτρα σε σχέση με την κυβέρνηση, αλλά ξέρουμε πόσο δύσκολο ήταν και σε σχέση με την προεδρική διακήρυξη και είναι ένα βήμα προς τα εμπρός και με ιδιαίτερη χαρά βρίσκω ότι διαβάζοντας παραγράφους 5 και 6 υπάρχουν αναφορές τώρα σε διασυνοριακές δράσεις η πρώτη φορά που έγινε δεκτό αυτό από την πενταμερή, τους Ρώσους και τους Κινέζους, να γίνεται λόγος για διασυνοριακές τέτοιες πρωτοβουλίες και δράσεις. Και αυτό μας νομιμοποιεί για τις κάποιες από τις δράσεις που είχαμε αναλάβει. Αλλά κάπως τις κάναμε υπό το ραντάρ, δηλαδή εισάγοντας ε, από την Τουρκία τέτοια αγαθά και διανέμοντας αυτά τα αγαθά σε περιοχές που δεν ελέγχονται από την κυβέρνηση. Εν πάση περιπτώσει, κάπως ανακουφίζει αυτό προς αυτή την κατεύθυνση και θέλω να αποτίσω φόρο τιμή στους ε, Λουξεμβούργιους φίλους διότι ήταν επικεφαλή σε σχέση με αυτό το ψήφισμα εκείνη με τους Αυστραλούς και μας ενημέρωναν πάντα ε, εκ του σύνεγγης για τα κείμενα αυτά και την προσπάθεια αυτή αλλά ήταν πραγματικά μια συλλογική προσπάθεια από όλους όσους εμπλεκόντουσαν και ενεπλάκησαν σε αυτό. Τώρα, λιγότερο ε, ανακουφιστικό είναι και αυτό αφορά και το, ένα τμήμα του, ψηφ, του ψηφίσματος τι θα γίνει με τις υποπολιορκία περιοχές ε, για παράδειγμα Χόμς, ε, Γιάμου και κάποιες άλλες περιοχές εδώ λοιπόν τι συμβαίνει βρισκόμαστε σε πραγματικά πάρα πολύ ευαίσθητο πεδίο για την πρόσβαση ιδιαίτερα σε σχέση με την ε, ε, αποχώρηση των γυναικών και των παιδιών και κάποιων από τους ε, άνδρες ή που φυλακίζονται και υποβάλλονται σε ανακρίσεις και για αυτούς που προέρχονται από το Χόμς πολλούς από αυτούς δεν ξέρουμε καν που βρίσκονται. Μπορείτε να φανταστείτε ποιες είναι οι υποθέσεις, οι εικασίες μας, ότι θα μπορούσε να συμβεί, να έχει συμβεί σε αυτούς. Είναι κάτι το οποίο παρακολουθούμε πάρα πολύ εκ του Διότι σε σχέση με την ανθρωπιστική δράση, όταν θέλουμε να προχωρήσει και βλέπουμε ότι το αντίθετο συμβαίνει, φυλακίζονται, βασανίζονται σε κρατητήρια και πρέπει εδώ να δούμε και σε σχέση με την ICC ε, μας αναφέρθηκε ότι να μην εκφράσετε ικανοποίηση υπερβολικά νωρίς διότι είναι πάρα πολύ ε, φρικαλέα η κατάσταση εκεί έτσι όπως συνεχίζεται. Στο ψήφισμα λοιπόν των Ηνωμένων Εθνών και σε σχέση με την ανθρωπιστική κοινότητα που καταβάλει προσπάθειες έχουμε μια δυνατότητα δράσης ε, για να δούμε ποια συνέχεια θα δίνεται και σε σχέση με τη Γενέβη και τη συνάντηση των υψηλών αξιωματούχων θα ήθελα απλά να πω ότι αυτό είναι κάτι που εμείς προσπαθήσαμε να προχωρήσουμε, να προαγάγουμε από πλευράς των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Όχι μόνο να υπάρχει αυτή η ομάδα υψηλών αξιωματούχων, αλλά να υπάρξει και αυτό το φόρουμ το φόρουμ για τη Συρία και όταν ε, ε, αυτό δεν προχώρησε όπως θέλαμε ε, μπορέσαμε να το προχωρήσουμε σε μια υψηλή ομάδα, ομάδα υψηλών αξιωματούχων Έχουμε τους Ιρανούς, ε, τους Σαουδάραβες, ε, τους ε, εκπροσώπους του Κατάρ και Πιστεύω ότι αυτό είναι επικοδομητικό να συμμετέχουν ώστε να γίνεται συζήτηση για τα θέματα πρόσβασης και προσπελασιμότητας και έχω κάπως την εντύπωση ότι αυτά όλα βοήθησαν στο να δημιουργηθεί ένα κλίμα αρρωγής και υποστήριξης για αυτό το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών στο οποίο καταλήξαμε και προχώρησε. Υπάρχει λοιπόν αυτή η συνάντηση στη Γενέβη πρώτη μετά από την έγκριση του ψηφίσματος. Η ιδέα είναι να ε, μπορέσουν οι επτά ομάδες εργασίας ε, που ε, καταρτίστηκαν να μπορέσουν να συνεχίσουν το έργο τους για τις πολιορκημένες περιοχές, για την ιατρική περίθαλψη και ιατρική φροντίδα. Να δούμε ποια πρόοδο σημειώνεται στους διαφορετικούς τομείς με αυτές τις πρωτοβουλίες μας. Κάτι άλλο, μια άλλη πτυχή σε όλα αυτά, ποια είναι είναι το ότι συνεχίζουμε να ασκούμε πίεση σε σχέση με όσους εμπλέκονται στο ανθρωπιστικό επίπεδο, να διασφαλίσουμε ότι αυτό το τελικό αποτέλεσμα θα είναι αποτελεσματικό σε σχέση με το κόστος που επενδύεται, κόστος όφελος, τι γίνεται εντός Συρίας, εκτός Συρίας, τι γίνεται στον κοινωνικό τομέα, τι γίνεται για την παιδεία, εκπαίδευση, κατάρτιση, για τα θέματα υγείας και την υγειονομική περίθαλψη. Όλοι θα πρέπει να συμμετέχουν σε μια επικοδομητική πολιτική ανοικοδόμησης ε, και ε, ε, δυνατότητας ανέγερσης της Συρίας που θα συγκλίνουν οι δράστες στο ανθρωπιστικό επίπεδο και στο επίπεδο της ανάπτυξης σε ένα κοινό επίπεδο σφαιρικό, ολοκληρωμένο, ολιστικά γιατί, διότι για παράδειγμα σε ένα στρατόπεδο μπορεί να υπάρχουν προγράμματα εκπαίδευση ή παιδεία και μπορεί να δει κανεί ότι αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα δαπανηρό. Να μην χρησιμοποιούνται λοιπόν ανθρωπιστικά κονδύλια αλλά να χρησιμοποιούνται κονδύλια για την ανάπτυξη ώστε να μπορούν αυτε οι δρασει να καλύπτονται. Ώστε όχι μόνο να υπάρχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα αλλά και καλύτερη εκπαίδευση και κατάρτιση για τα παιδιά. Και έτσι έμεσα και μπορεί να βοηθούν και άμεσα οι τοπικέ στον Λίβανο για παράδειγμα που είχε μια τεράστια εισρωή ε, προσφύγων ε, και που ήταν πάρα πολύ πάρα πολλές οι δυσκολίες ε, και που δόθηκαν τα κονδύλια τα περισσότερα υπέρ των προσφύγων αλλά καμιά φορά αγνοούμε, αμελούμε τις τοπικές κοινότητες κάπως και χρειάζεται μια ολοκληρωμένη σφαιρική, ολιστική στρατηγική που θα μεριμνά όχι μόνο για τους πρόσφυγες αλλά και για τις τοπικές κοινότητες. Χρειάζεται λοιπόν αυτή η δυνατότητα ε, ε, αλληλεμπλοκής θα έλεγα. Και Τέλος, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αδειμονώ να ξαναρχίσει η εκπροσώπησή μας, τα γραφεία μας ε, στη Δαμασκό. Πήρε επιτέλους ο συνεργάτης μας θεώρηση διαβατηρίου για να μπορέσει να εγκατασταθεί και να εργαστεί εκεί. Είναι σημαντικό να έχουμε εκπροσώπους επιτόπου εκεί, να είμαστε άμεσα σε επαφή επιτόπου με το τι τεκταίνεται και συμβαίνει εκεί με την παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκεί και ελπίζω ότι θα έχω καλές ειδήσει να σας διαβιβάσω προσεχώς. Και τώρα ε, εντάχει στρεφόμενος προς την κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία το επόμενο θέμα. Και πάλι χωρίς να υπερβάλλουμε εδώ υπάρχουν μικρές καλές ειδήσει, πολύ μικρές αλλά θετικές ειδήσει. Ο συνολικός αριθμός των εσωτερικά εκτοπισμένων μειώθηκε κατά τις τελευταίες πρόσφατες εβδομάδες ε, από 930 σε, ε, από 930.000 σε 700.000 αλλά ουσιαστικά αυτό μπορεί να εξηγηθεί αποκλειστικά με το ότι μετακινήθηκαν προς τον Μπαγκή, επέστρεψαν εκεί πάμπολοι. Έχουμε πάρα πολλούς όμως εσωτερικά εκτοπισμένους ε, στις επαρχίες και αυτό είναι εκείνο το οποίο με ανησυχεί περισσότερο γιατί δεν έχουμε και πολλές πληροφορίες ε, από αυτές τις ε, επαρχίες τι συμβαίνει με αυτά τα άτομα και τι ακριβώς γίνεται. Θέλω στους γιατρούς χωρίς σύνορα να αποτίσω φόρο τιμής και στην Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, διότι εκείνοι είναι, εκείνοι που προσπάθησαν να διατηρήσουν την εκπροσώπησή τους, τα στελέχη τους επιτόπου και να δούμε ότι τα στοιχεία τα οποία συλλέγονται δεν είναι πλήρη και υπάρχουν κενά. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία που μας δημιουργεί αυτό. Η επόμενη ανησυχία είναι ότι η κύρια αρτηρία από το Καμερούν δεν έχει ασφάλιση, δεν, έχει, δεν την χάνει ε, μ, περιβάλλοντος ασφάλειας. Αν πάει κανείς μόνος του με ένα φορτηγό υπάρχει κίνδυνος. Γι' αυτό υπάρχουν αυτοκινητοπομπές. Ε, ποιος είναι εκείνος ο οποίος θα παρέχει όμως την ασφάλεια ασφάλεια. Οι ένοπλες δυνάμεις sur le επιτόπου δεν μπορούν να καλύψουν όλες αυτές τις ανάγκες στον όγκο τον μεταφορικό που απαιτείται. Το να μπορέσουν λοιπόν να έρθουν ε, αυτοκινητοπομπές με ανεφοδιασμό είναι πολύ δύσκολο και το να μετακινείται κανείς με ελικόπτερα και πάλι εδώ πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι πάρα πολύ δαπανηρό και δημιουργεί προβλήματα. Τώρα ξαφνικά το 50% των κονδυλίων που μας δίνεται δεν θα ήθελα να παρεκτρέπονται ώστε να μισθώνονται και να ε, καλύπτονται ανάγκες για χρήση ελικοπτέρων. Θα θέλαμε άμεσα να χρησιμοποιηθούν για να παρασχεθεί άμεση βοήθεια ανθρωπιστική προς τους πληττόμενους. Όταν ε, ήρθα σε επαφή με την Επιτροπή Πιεσή του Συμβουλίου πρόσφατα τις προάλλες του είπα ότι δεν συμβαίνει πάρα πολύ συχνά να ακούει κανείς από τους ε, ανθρωπιστικούς ε, ε, από τα στελέχη ανθρωπιστικών υπηρεσιών κάτι τέτοιο αλλά έχουν πάρα πολύ, πολλές δυσκολίες να αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα προβλήματα και αναφέρθηκε και είπαμε ότι παρακαλούμε να υπάρχει μια δυνατότητα διασφάλισης ε, των εφοδιοπομπών διότι αν δεν υπάρξει διασφάλιση αυτής της συνιστώσας ασφάλειας δεν μπορούν να διοχετευτούν αυτά τα αγαθά στους ε, πληττόμενους πληθυσμούς και δεν μπορούμε να κάνουμε το έργο μας όπως πρέπει αφού γράστηκαν και άκουσαν ε, προσεκτικά συνεχίζουν τη μάχη που δίνουν ώστε να υπάρξει η δυνατότητα να διασφαλιστούν οι ενασχύσεις, οι ενισχύσεις που χρειάζονται, ευελπιστώ ότι θα μπορέσουν όλα να λειτουργήσουν με το σωστό τρόπο σε ένα μήνα, το πολύ σε δύο. Και αυτό θα ανακουφίσει κάπως την πίεση που υφίστανται οι γαλλικές ενόπλες δυνάμεις για να καλύψουν όλες αυτές τι ανάγκες. Είχαμε καλές ε, σχέσεις με τον ε, στρατηγό, είχα αρκετές συναντήσεις μαζί του και, του, ε, και δόθηκε και το παράδειγμα της Operation Serval στο Μαλί, όπου ο στρατιωτικό συντονισμό λειτουργήσε καλά και προ ήταν σε ένα πολύ διάφανο και ανοιχτό αποτελεσματικό πλαίσιο. Φυσικά προσπαθούμε οι ρόλοι να διαχωρίζονται και να είναι σαφείς, ώστε να υπάρχει η αμεροληψία και ουδετερότητα που πρέπει να διασφαλίζεται. Απαιτείται όμως αυτού του είδους η επαφή και ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων και ελπίζω πραγματικά ότι ο στρατηγός θα τα καταφέρει πρώτον να έχει τους πόρους και ε, τα, το, τα αναγκαία στοιχεία με τα οποία θα μπορέσει να δράσει ώστε να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια. Ε, είχα προαναφέρει και αν δει κανείς ένα χάρτη την εικόνα πως έχει. Θα δει κανείς ότι την κεντρική, κεντροαφρικανική δημοκρατία και αν φανταστεί κανείς ότι μπορεί να εξαφανιστεί σε μια μαύρη τρύπα αν δεν υπάρξει ασφάλεια, τότε αυτό θα έχει πραγματικά ε, ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις σε σχέση με την κατάσταση που είναι ήδη προβληματική σήμερα. Έχουμε μια μεγάλη πρόκληση στρατηγικού χαρακτήρα για τη διεθνή κοινότητα να αποκατασταθεί η σταθερότητα σε αυτή τη χώρα και αν μου επιτρέπετε να αναφέρω το εξής, αν δει ε, όλη την προσοχή που στρέφεται στο Κίεβο και την Ουκρανία κάπως θα με ανησυχούσε ότι θα ξεχνούσαμε ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλα σημαντικά κέντρα, φλεγόμενα κέντρα, Συρία, Μάλι, ε, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Σουδάν και ελπίζω να μην αμεληθούν αυτά και τα αγνοήσουμε και εστιαστούμε αλλού διότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να στρέφουμε την προσοχή μας ε, στις φλεγόμενες αυτές περιοχές ε, τα καλά νέα είναι ότι πρέπει να προσθέσω και να πω ότι χάρη στη δράση των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρία Στρίφλερ εσείς συμμετείχατε σε κάποιες από τις συνεδριάσεις και συναντήσεις που ε, διοργανώσαμε δίνοντας, ευαισθητοποιώντας για την κατάσταση στην κεντροαφρικανική δημοκρατία. Αυτό οδήγησε πολύ, σε πολύ μεγάλη αύξηση της βοήθειας από την Γαλλία προς αυτή τη χώρα. Το 2012 νομίζω 100 εκατομμύρια είχαμε από τη διεθνή κοινότητα διπλασιάστηκε αυτό το ποσό το 2013 και αυτό σε μεγάλο βαθμό χάρη στις δράσεις και τον ευδιάκριτο χαρακτήρα που δώσαμε σε αυτές τις πρωτοβουλίες. Καμιά φορά δεν επαρκεί να έχουμε μόνο μια σωστή ανάλυση των πραγματών. Πρέπει να διαχέουμε προς τα έξω αυτά τα στοιχεία, να διασφαλίζεται η υποστήριξη των φορολογουμένων και των αρχών στα διάφορα κράτη-μέλη. Επίσης ενεργοποιηθήκαμε ιδιαίτερα σε σχέση με τους Αμερικανούς, τους Καναδούς και να αποτίσω φόρο τιμή, τιμής και στους Βρετανούς οι οποίοι ενώ απουσίαζαν αρχικά ε, στη συνέχεια με πολλά κονδύλια ε, συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια για την κεντροαφρικανική δημοκρατία και αυτό μας κάνει να ευελπιστούμε για το μέλλον. Ένα σημαντικό στοιχείο πρόεδρε το αναφέρατε αυτό μια πολύ μεγάλη πρόκληση που εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε και συνδέεται με το θέμα της ασφάλειας είναι ότι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η ε, γεωργοί θα πρέπει να μπορέσουν ε, να καλλιεργήσουν και να, να, να μαζέψουν τον καρπό τους πριν από την ε, περίοδο των βροχών διότι διαφορετικά μπορεί να υπάρξει περίπτωση λιμού και να λιμοκτονούν μετά οι πληθυσμοί εκεί. Το ίδιο και για το Σουδάν. Οι εκτοπισμένοι άνθρωποι μακριά από τα χωριά τους χωρίς να έχουν πρόσβαση σε σπόρους και δυνατότητα να φυτέψουν, να καλλιεργήσουν πραγματικά βρίσκονται σε πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Ακόμα και αν υπάρχουν κάποια τρόφιμα τώρα, στο μέλλον θα σπανίζουν και θα εξαφανιστούν. Είναι πολύ σοβαρή αυτή η προοπτική. Να δοθεί λοιπόν, να δοθούν ε, σπόροι, αλλά χρειάζεται κυρίως ένα περιβάλλον ασφάλειας, να μπορούν να επιστρέψουν αυτοί στα χωράφια τους, να φυτέψουν τους σπόρους ε, και να δρέψουν τους καρπούς. Και για την ε, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία είναι η πρώτη φορά που η ΕΚΟ, η ανθρωπιστική βοήθεια τη Ευρωπαϊκή. Ένωσης ε, δίνει τη δυνατότητα από τον τομέα πολιτικής προστασίας ε, να καλυφθεί αυτή η ε, συνιστόσα. Πολλές φορές έχουμε συζητήσει για συνέργειες στο Ευρωκοινοβούλιο. Εδώ είδαμε ότι σε σχέση με την επιμελητία, χρησιμοποιώντας το πλαίσιο για την επιμελητία, αυξήσαμε το μεταφορικό δυναμικό, όχι με ελικόπτερα αποκλειστικά, αλλά με δυνατότητα με αεροσκάφη. Διάφοροι που δρούν εκεί μπορούν μπορούν να μεταφέρουν σε, με ένα κοινό φορτίο, με μία μεταφορά σε ένα αεροπλάνο, πιο αποτελεσματικά από πλευράς κομίστρου ή μισθώματος ε, ε, συγκεκριμένα φορτία σε αυτούς που έχουν ανάγκη να ε, ωφεληθούν από αυτά. Δύο λόγια για τον Νότιο Σουδάν τώρα, αν μου επιτρέπετε. Και το είχα προαναφέρει αυτό και κάποια άλλη φορά. Είναι μια κρίση πάνω και πέρα από την κατάσταση που ήταν κατάσταση κρίσης ήδη στο Σουδάν, αυτό το οποίο συμβαίνει στο Νότιο Σουδάν τώρα. Το είχαμε πει και το επαναλαμβάνω. Κάτι πήγε στραβά πολύ στραβά και γιατί δεν το προβλέψαμε. Γιατί δεν είμαστε προετοιμασμένοι έχοντας πάρει τα μηνύματα έγκαιρα όταν είχαμε την ανατροπή από την κυβέρνηση πέρσι το καλοκαίρι του ε, αρμόδιου γιατί δεν είμαστε ευφυείς να αντιληφθούμε ότι αυτή ήταν η συνταγή της καταστροφής των περιπλοκών που θα ακολουθούσε διότι ανήκουν σε διαφορετικές φυλές αυτοί οι δύο ε, εκείνος που αποχώρησε και εκείνος που τον ανέτρεψε. Και αν δεν υπάρχει δυνατότητα συμφιλίωσης ή συμβιβασμού, τότε αυτό μπορεί να οδηγήσει σε έκρηθμη κατάσταση και τεράστια προβλήματα. Πώς μπορεί να βελτιωθεί λοιπόν ο μηχανισμός μας πρόγνωσης κρίσεων, προ, πρόβλεψης και ε, κρίσεων. Τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να βελτιωθούμε και να έχουμε καλύτερες επιδόσεις. Νομίζω θα πρέπει να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Στο μεσοδιάστημα τα πράγματα είναι πραγματικά πάρα πολύ αρνητικά εντωμεταξύ. 900.000 εσωτερικά εκτοπισμένοι βρίσκονται σε αυτή τη χώρα. Έχει σταθεροποιηθεί κάπως αυτός ο αριθμός, αλλά όλο και περισσότεροι πρόσφυγες ε, καταφεύγουν στην Ουγγάντα... και βρίσκονται επίσης και στην ε, Αιθιοπία. Τα κονδύλια που δαπανούμε τώρα κατακαιρματίζονται. Το μεγαλύτερο μέρος καταλήγει στο Νότιο Σουδάν, αλλά υποστηρίζουμε, βοηθούμε και τους πρόσφυγες στις γειτονικές χώρες. Και πάλι σε αυτό πρέπει να πω ότι αν δεν φυτέψουν τους σπόρους και καλλιεργήσουν, είναι μια κατάσταση που δεν θα μπορέσουμε να την αντιμετωπίσουμε μετά την περίοδο των βροχών αν δεν γίνουν όλα όπως πρέπει να γίνουν και θα είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί μετά η κατάσταση αυτή διότι δεν θα υπάρχει το δυναμικό να υπάρχει η δυνατότητα διάθεσης τροφίμων. Δεν έχουμε αυτό το δυναμικό να διαθέσουμε όλα αυτά τα τρόφιμα. Είναι κάτι πάρα πολύ ανησυχητικό λοιπόν αυτό το οποίο μας αναμένει και το οποίο μεσοπρόθεσμα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Προσπαθούμε εκ προημίου να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε όσο το δυνατόν πιο νωρίς ε, δίνοντας προκαταβολές και ε, διασφαλίζοντας τα κονδύλια που χρειάζονται έγκαιρα για τον Νότιο ε, Σουδάν και στην ε, Επιτροπή μας, στην Επιτροπή θα γίνει συζήτηση και με τον κύριο Λεβαντόφσκι και με τον δικό μου ε, προϊστάμενο. Κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να προκαταβάλουμε χρήματα για να διασφαλιστούν όλες αυτές οι δράσεις όπως πρέπει. Και πιστεύω ότι το πολύ ανησυχητικό τελευταίο στοιχείο ως είδηση από τον Νότιο Σουδάν αλλά και πάλι δεν μπορεί να τους ε, ε κατηγορήσει κανείς είναι ότι ο Ρικ Ματσάρ ανέκτησε ε, μια συγκεκριμένη περιοχή το οποίο σημαίνει ότι η ροή πετρελαίου από την πολιτεία Unity θα πάψει να ε, μεταφέρεται, να διοχετεύεται και δεν θα υπάρχει τρόπος να επιστρέψει ανακάμψει η διεθνής κοινότητα και να αποκαταστήσει την κατάσταση πραγμάτων. Εδώ υπάρχει σαφής ε, επισήμαση και ένδειξη ότι η ασφάλεια, η συνιστόσα της ασφάλειας ε, έχει τεράστιες επιπτώσεις και τεράστια εμβέλεια ε, για τα θέματα της ανθρωπιστικής βοήθειας και των όσων μπορεί να κάνει η κοινότητα των χορηγών. Και πρέπει εδώ να πω ότι σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις για την ε, ειρήνη δεν είναι καλά τα μαντάτα. Δεν θέλουν ε, να διαβουλευτούν και να μπορέσουν να συμβιβαστούν μεταξύ τους οι αντίπαλοι δυστυχώς. Ολοκληρώνω και σταματώ εδώ πρόεδρε και είμαι πρόθυμος να απαντήσω σε οποιασδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια αν είναι δυνατόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Ντεγκεζέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη, κύριε Σόρνσεν, στην αρχή της ομιλίας σας απουσίαζα. Αν το έχετε καλύψει, παρακαλώ αγνοήστε την ερώτηση. Χαίρομαι καταρχάς πάρα πολύ και σας συγχαίρω και σας και το Γραφείο Ανθρωπιστικής Βοήθειας έχω για, το, για τη δουλειά που κάνετε στη Συρία. Χαίρομαι για τις χειορίσεις διαβατηρίων που καταφέρατε να επιτύχετε και αν ε, φτάσουμε μέχρι τη Δαμασκό είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε εκεί παρόντες. Εδώ στο ενημερωτικό σημείωμα που δώσατε για το ΕΚΟ και το ξεφίλησα λίγο, αναφέρεστε σε κάποιες περιορισμένες πρόοδους που έχουν ε, ε, επέλθει μετά τη δεύτερη διάσκεψη της Γενέβης. Βέβαια είναι κάπως ε, περιορισμένες αυτές οι πρόοδοι. Τι γίνεται ακριβώς στο Γιαρμούκ όμως σε σχέση με αυτό. Γιατί από ό,τι ακούμε άρχισε, σταμάτησε, ξανάρχισε, ξανασταμάτησε η βοήθεια. Αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε ακριβώς όταν πηγαίνετε στη Συρία, με ποιους συγκεκριμένους διάβλους εργάζεστε. Γιατί φαντάζομαι ότι δεν μπορείτε να κυκλοφορείτε παντού ελεύθερα στη χώρα. Έχετε διευρύνει αυτά τα κανάλια που είχατε δημιουργήσει με διάφορες ΜΚΟ ή ακόμα και την Ερυθρά Μισέλινο ε, καταφέρατε να διευρύνετε το πεδίο της δράσης σας ή απλώς έχει παραμείνει η κατάσταση ως ήταν και πώς συνεργάζεστε με το Συριακό Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων. Αυτό ήταν το πρώτο ερώτημα. Για τον Νότιο Σουδάν άκουσα πολύ προσεκτικά και έχετε δίκιο να εκφράζετε επιφυλάξεις για το γεγονός ότι όταν χρησιμοποιούμε ελικόπτερα τελικά πάνε χαμένα τα λεφτά της ανθρωπιστικής βοήθειας για ένα ε, μέσο μεταφοράς που είναι πάρα πολύ δαπανηρό. Στο Νότιο Σουδάν όμως δεν υπάρχουν υποδομές. Ε, πώς πάτε εκεί. Δηλαδή νομίζω ότι ακόμα και τα ψηφοδέλτια για τις εκλογές τα πήγαν με ελικόπτερο. Τώρα αυτή τη στιγμή έχετε δυνατότητες, έχει μέσα μεταφοράς που να είναι αρκετά αποτελεσματικά. Και ε, τι πιο πολιτική ερώτηση έρχομαι τώρα να κάνω. Στο Νότιο Σουδάν είναι πραγματικά ένας ε, αγώνας ε, εξουσίας μέχρι εσκάτων ε, και μετέρχονται όλα τα μέσα μέχρι και να διακινδυνεύσουν και να απειλήσουν ε, τη ροή του πετρελαίου εκεί που είναι η ίδια η πλουτοπαραγωγική πηγή της χώρας. Και δεν μπορεί κανείς από την ανθρωπιστική βοήθεια να συνεχίζει να χρηματοδοτεί αυτές τις ε, συγκρούσεις ε, για να καταλάβουν την εξουσία. Κάποια στιγμή θα πρέπει να καταλάβουν να έχουν ευθύνη αυτοί για τη χώρα τους. Ο Εμπέκη, νομίζω ήρθε στην Επιτροπή Εξωτερικών, δεν θυμάμαι ή εδώ, στην ΤΕΒΕ, ήταν σε ένα υψηλό πάνελ κατά της διαφοράς ο Μπέκη και τον ρώτησα κάτι για τον Νότιο Σουδάν για να δω τι κατάφερε να κάνει στο πάνελ και μας έλεγε ότι εντάξει μπορεί να είναι διαφορετικές εθνικές ομάδες, φυλές και τα λοιπά, αλλά δεν είναι ε, αυτή η αντιπαράθεση, είναι για την εξουσία και θα πρέπει η Ευρώπη να επιληφθεί και να λάβει υπόψη της και αυτό και όχι απλώς καλά πληρώνω τώρα και βλέπουμε ποιο ε, ε, είναι κατά την εκτίμησή σας τώρα το ε, καθεστώς που επικρατεί εκεί και τι γίνεται στη Συρία παρά την ημι αποτυχία της Γενέβης 2. Ευχαριστώ. Περνάει η ώρα, λέει η Πρόεδρος. Και νομίζω ότι θα ξαναδώσω το λόγο στον κύριο Σέρνσεν για να απαντήσει στις ερωτήσεις της κυρίας Ντέκεζε πριν τον ευχαριστήσουμε. Μάλιστα. Γνωρίζω ότι θα μπορούσαν να είχαν κάνει και πολλοί άλλοι ερωτήσει, αλλά πιέζει ο χρόνο. Να σα πω δύο λόγια για το Γιαρμόκ. Το πρώτο που ήθελα να θυμίσω, να πω αυτό που είπα και στην αρχή. Με ποιο τρόπο αντιμετωπίζουμε ε, όλες αυτές ε, τις ε, περιοχές που είναι υποπολιορκία. Κατά περίπτωση βγάζουμε κάποιους, ξαναβάζουμε κάποιους, τους στέλνουμε φυλακές. Αυτό είναι ε, περίπου ένα εργαλείο πολέμου από ε, τους αντιμαχόμενους. Εμείς που ασχολούμαστε με τα ανθρωπιστικά ε, νιώθουμε κάποια δυσφορία, αλλά όταν υπάρχει δυνατότητα μετάβασης τι να κάνουμε, μην πάμε. Αυτό συμβαίνει στο Γιαρμούκ. Η Ούνρα εκεί έχει πετύχει μια συμφωνία για να πάει, αν δεν απατώμε στις 26 Φεβρουαρίου πήγαν και έφεραν εφόδια, έβγαλαν και κόσμο από το Γιαρμούκ, αλλά τώρα Ε, έκλεισε και γίνονται και ανταλλαγέ πυρών, ε, θρικά πυρά, ε, με οβίδες, με ανταλλαγή πυροβολισμών και τα λοιπά. Ρουκέτες, δεν υπάρχει πρόσβαση πλέον. Και θα πρέπει να συνεχίσουμε όντως και έρχομαι στη συνεργασία μας. Πώς να το πω στο Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων είμαστε ευπρόσδεκτοι. Στη Δαυμασκό είναι άνθρωποι πάρα πολύ πολιτισμένοι, συζητάνε μαζί μας, μας εξηγούν κτλ. Εκεί που αρχίζουν να δυσκολεύουν τα πράγματα είναι όταν ερχόμαστε στις δυνάμεις ασφαλείας και ε, τις υπηρεσίες που ελέγχουν το στρατό. Γιατί χρειάζονται συνέχεια να κάνουν ελέγχους, διασταυρώσεις, λένε τη μία μέρα το ένα, την άλλη το άλλο, με επαλληνοδίες κτλ. Οι αρμόδιοι λοιπόν για την ανθρωπιστική βοήθεια είναι λίγο ε, ε, από από τα πραγματικά εμπόδια που υπάρχουν επί τόπου. Αυτό που εγώ ε, αντελήφθην μετά το Συμβούλιο Ασφαλείας είναι ότι οι θύνοντες, οι θύνοντες κατάλαβαν ότι έπρεπε να κάνουν κάποιες χειρονομίες. Ε, όπερ και γένετο, αλλά δεν ήταν αρκετό αυτό. Τώρα βλέπω μία πιστοχώρηση. Γιατί, γιατί έχει στραφεί η προσοχή αλλού τώρα όλων. Γιατί είναι πολύ λεπτά αυτά που γίνονται. Οι άνθρωποι δεν είναι αφελείς και μας χρησιμοποιούν κιόλας και παίζουν. Ε, ε, το ΣΑΚ είναι μια οργάνωση ανθρωπιστική που είναι η πιο ευρέως διαδεδομένη στην περιοχή. Και ε, ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός μας είπε ότι στο 90% των περιπτώσεων προσπαθούν να έχουν ανθρωπιστική δράση, κάνουν τεράστια δουλειά, έχουν και θύματα, σκοτώνονται οι δικοί τους. Δεν σημαίνει ότι είναι όλα ρόδινα. Αλλά παρόλα αυτά είναι το σημαντικότερο Ε, τους χρησιμοποιούν εκεί και τα Ηνωμένα Έθνη και η ΜΚΟ. Ναι, στη διαφοροποίηση ναι, ε, διευρύναμε το ε, φάσμα των ΜΚΟ που λαμβάνουν κοινοτική χρηματοδότηση, ιδιαίτερα για τη διασυνοριακή. Άλλαξε λίγο η γλώσσα, γιατί τώρα μπορώ να, το λέω. Στο παρελθόν λέγαμε ότι θα πρέπει με κάθε τρόπο να έχουμε πρόσβαση. Αυτό είναι εφημισμός. Δηλαδή, κάθε τρόπο σημαίνει ότι περνά στα σύνορα μια κυρίαρχη χώρα χωρί να τη ρωτήσει. Ε, τώρα μετά το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών έχουμε ξεκαθαρίσει και τη γλώσσα μας και κατάλαβε και, και η Συριακή κυβέρνηση πλέον ότι θα πρέπει να το δεχτεί. ότι συμβαίνουν αυτά. Ε, πάντως σίγουρα δεν είναι επαρκή όσα συμβαίνουν. Θα πρέπει να εξακολουθήσουμε να πιέζουμε και μπορεί τώρα με τους Ρώσους κάπου για άλλα θέματα να συγκρουόμαστε. Ε, ο διάλογος πρέπει να παραμένει ανοιχτός γιατί χωρίς τους Ρώσους αποκλείεται να βελτιωθεί και η κατάσταση. Με κάποιο τρόπο πρέπει να συνεργαστούμε. Για τον Νότιο Σουδάν συμφωνούμε. Τα ελικόπτερα ε, κοστίζουν ε, του κόσμου τα λεφτά. Ο Κούκος Αϊδόνη ε, και αν αρχίζω να πληρώνω ελικόπτερα πάει ο προϋπολογισμός. Στο παρελθόν μπορούσαμε να φέρνουμε ε, με βάρκες σε ένα νησί ε, τρόφιμα και εφόδια. Υπάρχουν και φορτηγά, αλλά όλα σταματάνε όταν αρχίζουν οι βροχές. Οπότε μόνο εναέρια μέσα, ελικόπτερα και αεροπλάνα βοηθούν. Και θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε, θα δούμε τι λεφτά θα έχουμε τότε στο γκουμπάρα μας. Ε, τώρα, για την μάχη για την εξουσία που είπατε, έχετε δίκιο. Ε, δεν είναι μεταξύ φυλών εκεί οι διενέξεις και οι σύραξεις. όχι. Ε, πρόκειται για πρόσωπα που θέλουν να καταλάβουν την εξουσία. Αλλά στο δρόμο για την εξουσία κάνουν κάποια λάθη που μετά έρχονται να διχάσουν τις φυλές. Και τώρα υπάρχει ε, ε, διχασμός ανάμεσα στις φυλές στο Νότιο Σουδάν. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θέλω να ρίξω λάδι στη φωτιά. Σας περιγράφω ότι ισχύει. Ε, έχει εκφυλιστεί κάπως η κατάσταση και ακολουθεί και τα όρια των φυλών και τις φαίνει αντιμέτωπε, και τι μπορούμε να κάνουμε για να ξαναγυρίσουμε στην αρχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέτε θα πρέπει να διαστηριοποιηθεί, ε, όχι μόνο και οι Αμερικανοί, όλοι οι μεγάλοι. Θυμάμαι την πρώτη φορά που πήγα στην Τζούμπα, μίλησα με την Αμερικανίδα πρέσβερ και της είπα ότι κοιτάξτε μήπως να συνεργαστούμε. Και εδώ αυτοί που είναι στην κυβέρνηση δεν είναι τίποτα γελούδια. Αλλά μετά την ανεξαρτησία κυριαρχούσε αυτή η ιδέα ότι ε, πολέμησαν τόσο πολύ με το Σουδάν, τώρα είμαστε όλοι αισιόδοξοι και θα χτίσουν τη χώρα τους, αλλά δεν είχαμε δει ότι δεν είναι εύκολο έναν αντάρτη να τον κάνεις ε, δημόσιο υπάλληλο. Ευχαριστώ κύριε Σόρενσεν που μας ήρθατε να μοιραστείτε μαζί μας ε, όλη αυτή τη δουλειά της ΕΚΟ στην κρίση και κινδυνεύει να έρθει να προσθεθεί άλλη μια ανθρωπιστική κρίση και όταν τα σκέφτομαι αυτά πραγματικά τρομάζω σκεπτόμενοι και το δικό σας προσωπικό και την ε, υγεία του μεταξύ άλλων. Ευχαριστώ πολύ και ε, να ξέρετε ότι θα παρακολουθούμε πολύ στενά τις εξελίξεις και το γεγονός ότι να έχετε, θα φροντίσουμε να έχετε χρήματα. Ευχαριστώ, λέει ο κύριο Σόρεσεν. Να μην πέστε θύματα ε, στις άτυχες ε, περικοπές του προϋπολογισμού. Αύριο έχουμε κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Προπολογισμών για τη χρηματοδότηση ανθρωπιστική βοήθεια. Το λέω αυτό προ τα μέλη τη Επιτροπή μα για να μεταβείτε εκεί. Σας ευχαριστώ. Τώρα έχουμε ψηφοφορίες. Να πάτε στο καλό. Αρχίζει η ψηφοφορία. Βγάλτε τις κάρτες.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 του ελεγκτικού συνεδρίου σχετικά με τη στήριξη της Ένωσης στη διακυβέρνηση λαϊκής δημοκρατίας του Κονγκό. Πρώτα θα ψηφίσουμε τις ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης. Χωρίς τροπολογίες. Ψήφι υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Ensuite, la question à la Commission qui est pour... στην Επιτροπή, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Okay. Ε, ο κύριος Μίτσελ, υπάρχει δυνατότητα να μην ψηφίσουμε την επόμενη, ρωτάω. Ε, να ψηφίσουμε unblock, συγγνώμη, όλα μαζί τα υπόλοιπα. Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Η τροπολογία είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 10 υπέρ κατά απόχες απορρίπτεται. Η τροπολογία 11 ειπέ κατά απόχες απορρίπτεται. Η τροπολογία 12 ειπέ κατά απόχες εγκρίνεται. Η τροπολογία 13 υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται. Η τροπολογία 14 ειπέ κατά απόχες απορρίπτεται. 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 17 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 18 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Η τροπολογία 1 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 3 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 4 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 6 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 7 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα το σύνολο του ψηφίσματος όπως τροποποιήθηκε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και η ηλεκτρονική ψηφοφορία αρχίζει τώρα για καλό και για κακό. Πέρασε. Ομόφωνα. Εγκρίθηκε. Θαυμάσια. Άλλο. Nous, nous ε, τώρα θα ψηφίσουμε το κείμενο που αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης από τον κύριο Γκέρνς για την απόφαση να υπάρξει Ευρωπαϊκό έτος ανάπτυξης, λέει εδώ. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Et vote électronique, le vote est η ηλεκτρονική επαλήθευση αρχίζει ναι. τώρα. Ένας. Ομόφωνα επίσης εγκρίθηκε. Alors, euh, nous votons sur la recommandation. Ψηφίζουμε τώρα για τη σύσταση προς το Συμβούλιο σχετικά με την ανθρωπιστική δράση μη κρατικών δυνάμεων με σκοπό την προστασία των παιδιών. Είναι η έκθεση της κυρίας, κυρίας Αρχεντίνη. Η τροπολογία 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Έχουμε εδώ προφορική τροπολογία παριθμών 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Επόμενη καταπίπτει, οπότε... Έχουμε τροπολογία 5, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η προφορική τροπολογία υπαριθμών 2, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η συγγήτρια. Τα υπόλοιπα μπορούμε να τα ψηφίσουμε όλα μαζί. Δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε. Καλά, δεν πειράζει. Η τροπολογία 7 υπέρ. Εγκρίνεται. Η 8 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα, έχουμε την τροπολογία 10 τώρα σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα θα ψηφίσουμε το σύνολο, όπως τροποποιήθηκε, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος ε, ηλεκτρονικός αρχίζει τώρα. Πέρας. Ομόφωνα επίσης. Υπερψηφίστηκε. Και μπράβο κύριε Σαρχεντίνη. Τώρα η έκθεση του κυρίου Αρσένη. Σύσταση προς το Συμβούλιο. Ένα υπέρ κατά αποχές Δύο υπέρ κατά Yes, απορρίπτεται. τρία σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά yes, εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ κατά yes, εγκρίνεται. Πέντε υπέρ κατά yes, απαρρίπτεται. τέσσερα υπέρ κατά χες απορρίπτεται 6 υπέρ κατά χε, εγκρίνεται 7 υπέρ κατά χες εγκρίνεται 8 υπέρ κατά χες εγκρίνεται 9 υπέρ κατά χες εγκρίνεται 10 υπέρ κατά χες εγκρίνεται το σύνολο της γνωμοδότησης υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ηλεκτρονικά τώρα ηλεκτρονικά ομόφωνα εγκρίθηκε Α, όχι, όχι ομόφωνα, δύσφωνα με τέσσερις ψήφους κατά, ετερόφωνα. Τώρα η έκθεση Γκέρινς για την συνέπεια της ανάπτυξης. Προφορική τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Χες. Εγκρίνεται. 9 υπέρ. Κατά. Χες. απορρίφτεται 10 υπέρ. Κατά. Χες. Εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά χες εγκρίνεται 12 όχι 13 υπέρ κατά <clears throat> από χες απορρίψεται συμβιβαστική α υπέρ κατά χες εγκρίνεται τροπολογία 15 υπέρ κατά χες απορρίπτεται. 16 υπέρ κατά χθες εγκρίνεται. 19 υπέρ <clears throat> κατά χθες εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά χες αν 21 υπέρ α όχι έχει καταπέσει 22 υπέρ κατά χες εγκρίνεται 23 δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά χες εγκρίνεται δεύτερο τμήμα δεύτερο τμήμα όχι, επαλήθευση για το πρώτο τμήμα ηλεκτρονικά. Πρώτο τμήμα 23. Μια έλεξη. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Χες εγκρίνεται. 24 υπέρ υπέρ, υπέρ, υπέρ, κατά. Εποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική Β υπέρ, κατά. Χες, εγκρίνεται. 29 <laughs> Υπέρ κατά αποχές απαρρίπτεται 30 υπέρ κατά αποχές απαρρίπτεται 31 υπέρ κατά αποχές απαρρίπτεται 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 33 υπέρ κατά χες Απορρίπτεται. 34 υπέρ κατά Α, όχι, 36, 36, καλά, 36, 36, 36 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, χες, απαρρίπτεται.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 35 υπέρ κατά αποχές απαρρίπτεται. Υπάρχει πρόβλημα σε, μερικές, ε, σε μερικούς καταλόγους ψηφοφορίας των πρασίνων. Λοιπόν, 35 ηλεκτρονικά. 35 ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία. Τι ψηφίζουμε λοιπόν. Το ξέχασα. 35. 35. Α, 35 γιατί δεν έχω το σωστό κατάλογο, καταλάβατε. 35. Δεν έχω το σωστό κατάλογο. Διαδικαστικό κυρία Πρόεδρε, εδώ υπάρχει μια σύγχυση. Κυρία Πρόεδρε, μπορώ να θέσω ένα διαδικαστικό. Υπάρχει μια σύγχυση. Τι έγινε με την τροπολογία 2, τι έγινε. Ε, όχι 37, 37, 37. Α, εγκρίθηκε, α, καλά, α, τότε καλά. So, is it 35? Oui. Le vote, donc le vote est toujours ouvert, on manque un vote. Sur l'amendement 30. Λοιπόν, για την 35 είπαμε, ηλεκτρονικά. Έλξε. Έλξε. Εγκρίνεται. Και D'accord. Donc, on a... Amendement oral. Non, non, non, non, on les vote, parce que donc, ça n'a pas été adopté. Tu, tu, tu, Et là, donc l'amendement oral 3, euh, qui, est, qui est en, en faveur Υπάρχει μια προφορική τροπολογία. Υπέρ, κατά, ποιες εγκρίνεται. Τριάντα τέσσερα υπέρ, κατά χέσαν απαρρίπτεται 38 υπέρ κατά χες εγκρίνεται η προφορική τροποποίηση λοιπόν τώρα των πρασίνων υπέρ τα χες εγκρίνεται Σαράνδα υπέρ κατά τες απαρρίπτεται ένα, υπέρ κατά χες απορρίπτεται δύο, υπέρ κατά χες απαρρίπτεται 43 υπέρ Καλά, πρόεδρε, πρόεδρε. Τι θέλετε για τη 42, επαλήθευση, ωραία. Για τη 42 επαλήθευση. Δεν έχω το σωστό κατάλογο. Δεν έχω το καλό, το σωστό κατάλογο. Λοιπόν, έληξε. Εγκρίνεται 43 υπέρ κατά χε απορρίπτεται. 1 υπέρ κατά χε εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά χε απαρρίπτεται 3 υπέρ τα εσ αγκρίνεται 4 και 5 υπέρ κατά εποχές εγκρίνονται 6 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται προφορική 4 υπέρ κατά και εγκρίνεται ίσως την 7, την 8 και την προφορική 5 όλες μαζί υπέρ, υπέρ, υπέρ μπλοκέ κατά αποχές εγκρίνονται τώρα το σύνολο όπως έχει τροποποιηθεί υπέρ κατά και εγκρίνεται και η ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται έληξε πανηγυρικά εγκρίθηκε Mais on a terminé. Pas de Τίποτα διάφορα έχετε? Όχι. Επόμενη συνεδρίαση 25 Μαρτίου 9 με 12.30 και 3 με 6.30 το απόγευμα. Τώρα θα συνεχίσουμε και κλεισμένον το θυρών της συνεδρίαση, όχι ότι τελειώσαμε. Ε, θα συζητήσουμε για το στρατηγικό διάλογο.